Buenas tardes a todos. Voy a presidir la sesión en Αγαπητοί συνάδελφοι, την 5η Σεπτεμβρίου του 2019 οι συντονιστές της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ συμφώνησαν ε, να οργανώσουν μια ανταλλαγή απόψεων ε, σε τούτη την Επιτροπή σχετικά με το πολύ ευαίσθητο θέμα των ε, παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, των ξένων μαχητών, καθώς επίσης και την ενδεχόμενη επιστροφή τους, επαναπατρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης αποφάσισαν να ε, ε, ε, καλέσουν τις υποεπιτροπές του ΑΚΕΣΕΝΤΕ να συζητήσουν από κοινού, οι επιτροπές λοιπόν έλεγαν του για το θέμα αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη είναι τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς επίσης και τις πολλαπλές υποθέσεις που έχουν φτάσει ενώπιον των δικαστηρίων διαφόρων κρατών μελών, που έχουν απαντηθεί αλλά που κυρίως ε, έχουν ε, δεχθεί διαφορετική ανταπόκριση ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να οργανώσουμε μια συζήτηση κατά την έννοια αυτή. Πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή εστίαση και ευρωπαϊκή λύση και ελπίζω εκ βάθους καρδίας ότι ότι αυτή η συζήτηση θα συμβάλλει ε, στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι ε, άνθρωποι. Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, τις Προέδρους κυρία Αρενά της Επιτροπής Δρουά καθώς επίσης και της κυρίας Λουαζό, Πρόεδρο της ΕΝΤΕ. Θα ήθελα να καλέσω θα καλέσω την κυρία Λουαζό να κάνει μια πρώτη σύντομη τοποθέτηση. Πριν, ε, μετά θα κάνουν ε, τις παρεμβάσεις τους οι καλεσμένοι μας και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις-απαντήσεις. Να σας πω επίσης ότι οι συγγενείς κάποιων από των παιδιών που φύγονται από την κατάσταση αυτή ε, βρίσκονται μεταξύ του ακροατηρίου ε, και τους ε, χαιρετίζω εξ ονόματος αυτής της Επιτροπής και τους καλωσορίζω στις συζητήσεις μας εδώ και πραγματικά εκ βάθους καρδίας επιθυμούμε αυτή η συζήτηση να έχει σαν αποτέλεσμα με πιο συντονισμένη ανταπόκριση της του θέματος. Έχουμε εδώ την κυρία Μαλίκα Μάλμη, την κυρία Μαγιάτ Μαρισούλ, τον κύριο Γρής Γκούταλη, την κυρία Σάρα Βερχόβεν, την κυρία Σαμίρα Λάκεν, την ε, κυρία Γιλτής Καραμάν, την κυρία Φατή Χαλαχά, την κυρία Ματιά Ροσαρόσο, την κυρία Γκίτα Μελχάχ και την κυρία Ναβίλα Μαθχούθ.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 και επαναλαμβάνω ότι ευχόμαστε βάθος καρδίας ε, την ε, βέλτιστη δυνατή επίλυση του προβλήματός σας. Ε, είναι εδώ μαζί μας η κυρία Ρενά και η κυρία Λουαζό. Θα δώσω πρώτα για δύο λεπτά τον λόγο στην κυρία Λουαζό και μετά στην κυρία Ρενά γιατί με αυτή τη σειρά με καθοδήγησε η γραμματεία να δώσω τον λόγο. Κυρία Λουαζό, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαϊτέ το θέμα που μας ε, απασχολεί σήμερα είναι ένα ε, ακαθόδες και αναπίτρεπτο ε, ζήτημα στα πλαίσια της τραγωδίας που εδώ και 8 χρόνια ζει η Συρία. Στο επίκεντρο αυτής της τραγωδίας έχουμε βεβαίως την, τραγική μοίρα των παιδιών της Συρίας, παιδιά τα οποία καθόλου δεν ευθύνονται για την τραγωδία που έχει πέσει πάνω τους. Ναι. και επίσης εντός του προβλήματος αυτού ε, υπάρχει το πρόβλημα των παιδιών των τζιχατιστών, ε, πολλά εκ των οποίων έχουν γεννηθεί στη Συρία όπου πήγαν να πολεμήσουν οι γονείς τους. Δεν ζήτησαν τίποτα όμως τα παιδιά αυτά. Ε, δεν θέλησαν τίποτα, δεν αποφάσισαν τίποτα, μόνο υφίστανται και ταλαιπωρούνται και υποφέρουν. Οι γονείς τους αποφάσισαν ε, να τους ε, ε, κάνουν να υπομείνουν όλες αυτές τις ταλαιπωρίες. Η ΝταΕΣ είναι αυτή που αποφάσισε να τους βάλει στο επίκεντρο αυτού του προβλήματος. Αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η ευθύνη μας. Θα τους αφήσουμε εκεί να σιγοπεθαίνουν στα στρατόπεδα. Ε, θα τους αφήσουμε να ταλαιπωρούνται μέσα σε φρικτές και ακατονόμαστες ταλαιπωρίες. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ήδη κάνει κάποιες προσπάθειες για να επαναπατρίσουν τα παιδιά αυτά και θα πρέπει να χαιρετήσουμε αυτές ε, τις προσπάθειες. Ωστόσο, ε, σκόνταψαν σε πολλές δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες θα πρέπει να γίνουν γνωστές γιατί η κατάσταση έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Ξέρουμε ότι πολλές γυναίκες στα στρατόπεδα δεν αφήνουν ε, τα παιδιά τους ε, να φύγουν. Η κατάσταση όμως στα στρατόπεδα γίνεται όλο και χειρότερη. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα παιδιά αυτά γιατί ούτως ή άλλως μια τέτοια κίνηση δεν θα βελτίωνε την ασφάλειά μας. Πρέπει να κινηθούμε και αυτό πριν είναι πολύ αργά. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λουαζό για όσα μας είπατε. Η κυρία Αρενά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε σε αυτήν την συζήτηση για τα παιδιά των ξένων μαχητών. Είναι ένα ζήτημα ε, ε, δύσκολο, ε, δυστυχώς γιατί ε, λυπηρός πολλές κυβερνήσεις δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα. Αλλά όπω είπε και η Νεταλή προηγουμένω, δεν μα οδηγεί σε ε, κανένα αποτέλεσμα το να ε, στρέφουμε το κεφάλι μα από την άλλη πλευρά. Μιλάμε για παιδιά, ε, των οποίων οι γονείς προφανώς εγκλημάτισαν, ωστόσο παραμένουν παιδιά, κυρίως παιδιά και κυρίως θύματα. Και ως θύματα θα πρέπει να χαίρουν προστασίας. Είναι πολλές ε, οι μελέτες ε, οι οποίες ε, συμπεραίνουν εν τέλει ότι το ψυχολογικό βάρος αυτών των παιδιών που έχουν ζήσει στον πόλεμο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα τους ακολουθήσει σε όλη τους τη ζωή. Ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα μοιραίο και δεν υπάρχει τίποτα αναπόφευκτο και μη αναστρέψιμο όταν μιλάμε για παιδιά. Παιδιά τα οποία αναλαμβάνουν ε, ε, από ε, έμπειρους ανθρώπους νωρίς μπορούν να ξεπεράσουν σιγά σιγά τα προβλήματα τα οποία έχουν αντιμετωπίσει, τις δυσχέρειες που έχουν ζήσει και επομένως να σπάσουν το φαύλο κύκλο της βίας. Στις 20 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει μία υψηλού επίπεδου συζήτηση για το θέμα αυτό. Υπάρχει μία σύμβαση η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Πρόκειται για μία σύμβαση για τους ανηλίκους που αναφέρει ότι πριν από τα 18 ένα παιδί θεωρείται παιδί, έχει δικαίωμα στη ζωή, έχει δικαίωμα στην προστασία της ταυτότητάς του, έχει το δικαίωμα να ζήσει με τους γονείς του αλλά και να ε, ε, ε, επανενωθεί με την οικογένειά του. Επίσης, είναι ε, ε, παιδί το οποίο θα πρέπει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ένωμη τάξη της χώρας του ε, και εάν αυτή προβλέπει πιο θετικά στοιχεία από την σύμβαση ε, να ε, ε, απολαμβάνει αυτών των δικαιωμάτων. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τα παιδιά των ξένων μαχητών. Είναι γεγονός ότι οι γονείς έκαναν εγκλήματα, αλλά θα πρέπει να μελετήσουμε, να δούμε τα παιδιά αυτά σαν παιδιά πριν μελετήσουμε τι γίνεται με τους ή τι έχουν κάνει οι γονείς τους. Βεβαίως γνωρίζουμε τους εκβιασμούς που ορισμένοι γονείς ασκούν λόγω των παιδιών. Εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να τολμήσουμε, δεν θα πρέπει να διστάσουμε. Ε, ας φέρουμε τους ανθρώπους αυτούς εδώ, ας τους δικάσουμε με τρόπο ε, δίκαιο. Πρέπει να πω ότι έχουμε και την κυρία Ανιέσα Καλανμάρ, η οποία ε, έχει ασχοληθεί με το θέμα. Εκείνη λοιπόν, η κυρία Καλαμάρ λέει ότι δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις. Ε, θα πρέπει ε, αυτοί οι ξένοι μαχητές να δικαστούν στις χώρες στις οποίες έχουν διαπράξει τα αδικήματα, γιατί θα πρέπει να δώσουν λύση, θα πρέπει να δικαστούν απέναντι στα θύματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις και εν συνεχεία το λόγο θα λάβουν οι συντονιστές και θα ακολουθήσουν ε, άλλοι βουλευτές από τη Λίμπη, από την Τροιά, τη που ενδιαφέρονται για το θέμα. Είναι περιορισμένος ο χρόνος, οπότε θα σας παρακαλούσα να δηλώσετε το συντομότερο δυνατό ήδη από τώρα στη Γραμματεία ΛΥΜΠΕ αν θέλετε το λόγο, οπότε έτσι θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε καλύτερα τους χρόνους. Και θα είμαι και άτεγκτη. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή με το χρόνο, εφόσον έχω υπολογίσει πόσα λεπτά θα έχει ο καθένας. Και σίγουρα όλοι έχετε να πείτε πολύ σημαντικά πράγματα. Ε, πρέπει να σεβαστούμε και το δικαίωμα του λόγου όλων και το δικαίωμα, ε, μάλλον και την παρουσία των προσκεκλημένων μας εδώ. Ε, ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρή Ντομινίκη Παγάου, που είναι υπεύθυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Περιφερειακού Γραφείου της ΥΠΑΤΣΕΙΣ Αρμοστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά και σας ευχαριστώ ήδη προκαταβολικά για την παρουσία σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που οργάνωσε την ανταλλαγή αυτή απόψεων και προσκάλεσε στην υπατερμοστή ε, για δικαιώματα στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω συντομία τι κάνει το γραφείο μας, ε, τι κάνει η υπηρεσία μας. Είμαστε ε, ενεργό μέλος του Συμφώνου για την Αντιτόπιση Τρομοκρατίας σε τομείς που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη, την πρόληψη βίας, εξτρεμισμού και ε, τη συμπερίληψη τη διάστασης του φίλου πολιτικές. Είμαστε στο, ε, στην ομάδα εργασίας για την προστασία κράτου δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θέλουμε να υπάρχει λογοδοσία αλλά και σεβασμός για τα δικαιώματα των θυμάτων. Επίσης είμαστε υπέρ μιας προληπτικής ε, προσέγγισης, έχουμε κατευθυντήρες γραμμές, σε σχέση και με τις απειλές ε, των ξενομαχητών, το βλέπετε αυτό το έγγραφο και έχουμε και πολλά άλλα φυλάδια. Θα σας στείλω τον ε, κατάλογο, συγκεκριμένα στην γραμματεία της Επιτροπής σας. Ε. Έχουμε ένα γραφείο στο, στη Βηρητό για τη Συρία και επίση. Ε, παρέχουν υπηρεσίες και στην υπηρεσία της Γενέβης για την κατάσταση της Συρίας. Ό,τι αφορά τώρα τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών, ε, δεσμευόμαστε από αυτή την ε, σύμβαση. Πρέπει να βοηθούμε τα παιδιά έως 18. Όλες οι δραστηριότητες των ξενομαχητών επηρεάζουν τα παιδιά, θύματα, μάρτυρες ε, ή ε, φέρουμε ως δράστες ενίοτε πολλές φορές ε, τα στρατολογούν ε, στο ίντερνετ και κάποια καταναγκαστικά, εξαναγκαστικά ως θύματα διακίνησης ή κάποια που τα φέρνουν κάποιες συγγενείς τους ή κάποιοι οποίοι, ε, κάποια που ζούσαν σε κατεχόμενα από το Ισλαμικό κράτος εδάφη. Πολλές φορές έχουμε παιδιά τα οποία έχουν κινηθεί από γονείς ξένους μαχητές, είτε και ο Θεόλος, είτε είναι αποτέλεσμα βιασμού. Αυτό που ζητούμε είναι ο επαναπατρισμό. Θα έχετε δει ίσω τη δήλωση τη Δευτέρα ε, του εκτελεστικού διευθυντή τη UNICEF. Ζητά από τι κυβερνήσει να επαναπατρίσουν τα παιδιά. Και αυτό προτούν αναργά. Επίσης, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Παιδιών του ΟΗΕ έχει συστήσει φέτος το Φεβρουάριο στο Βέλγιο να ε, διευκολύνει την επιστροφή, τον επαναπατρισμό των Βέλγων, ε, των οικογένειών και των παιδιών κυρίως. Το ίδιο κάνει και ο ειδικό απεσταλμένο ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σε διαβουλεύσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη το ίδιο έκανε ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επίτροπος, η οποία είπε ότι Πρέπει κατεπηγόντως να επαναπατριστούν ε, οι ξένοι και οι οικογένειές τους. Ε, γιατί αυτό είναι το μόνο σύνομο με το διεθνές δίκαιο. Η κατάσταση των παιδιών και των ενηλίκων ε, σίγουρα είναι πολύπλοκη και σε αυτά τα δέκα λεπτά που έχω θα ήθελα να εστιάσω σε τρία σημεία. Καταρχάς να σας κάνω ένα σύντομο απολογισμό της κατάστασης στη Συρία και Ιράκ. Δεύτερον, να μιλήσω για τις υποχρεώσεις των κυβερνήσεων απέναντι στα παιδιά είτε είναι ύποπτα είτε όχι για παραβίαση των δικαιωμάτων και τρίτον να σας μιλήσω για τις θεμητές ανησυχίες των κρατών μελών για τα θέματα της ασφάλειας και θα μιλήσω για αντιμετώπιση ή πρόληψη της τρομοκρατίας. Ξεκινώ με την κατάσταση επιτόπου. Φυσικά εδώ μιλάμε για παιδιά εγκλωβισμένα σε δύο χώρες που αντιμετωπίζουν δεινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της τρομοκρατίας. Στο Ιράκ Έχουμε σχεδόν 1,8 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπιστέντα άτομα και 6,7 εκατομμύρια άτομα τα οποία χρήζουν ανθρωπιστικής προστασίας. Προστασία, βοήθεια, αυτή είναι η προεξάρχουσα προτεραιότητα από ανθρωπιστικής πλευράς. Είναι περιορισμένες οι δυνατότητες όμως για εθελούσια και ασφαλή επιστροφή αυτών των ανθρώπων. Είδαμε και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις πρόσφατα της Τουρκίας που επιδίνωσαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση ε, και βλέπουμε ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες ε, οικογένειες να καταλείπουν ε, τη Σύρια και το Ιράκ. Στη Συρία έχουμε 10,7 εκατομμύρια ανθρώπους που πλήττονται από αυτή τη σύγκρουση. 5 εκατομμύρια σε αυτό είναι παιδιά. Κατάσταση στη Συρία πάρα πολύ ανησυχητική. 2 εκατομμύρια παιδιά στη βορειοανατολική Συρία πλήττεται πιο πολύ από το προηγούμενο έδαφος που σας ανέφερα της Συρίας. Έχουμε 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν ε, σε κατάσταση ε, τραγική και σε ό,τι αφορά τι Δημοκρατικές Δυνάμεις ε, έχουν ένα καταβλισμό με 70 περίπου χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά και γυναίκες από τις 70.000 είναι το 90%. Μιλάμε για πάρα πολλού εσωτερικά εξοπιστέντες ε, με τραϊκέ ε, συνθήκε διαβίωση και με τη στρατιωτική επέμβαση τη Τουρκία ε, και την έλευση του χειμώνα τα πράγματα επιδεινώνονται. Είναι δύσκολο να βρεθούν τα δεσμά με ξένου μαχητέ, οι δεσμοί των παιδιών με του ξένου μαθητέ. Με βάση εκτιμήσει τη UNICEF και άλλων και του Ινστιτούτου EGMON, υπάρχουν σχεδόν 28.000 παιδιά από 60 διαφορετικέ χώρε ή 16 δεν είναι σαφές από την ομιλήτρια και παραμένουν αυτά τα παιδιά σε καταβλισμού στο μεγαλύτερό τους ε, αριθμό και για τη Συρία ε, δεν έχουν καν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τους καταβλισμούς αυτούς. Ε, είναι σχεδόν κέντρα κράτηση. και λιγότερο από 20% των παιδιών αυτών είναι πάνω από 12 χρονών. Τα μισά είναι κάτω από 5 χρόνων. Και η τεράστια πλειοψηφία των παιδιών αυτών, τα 20.000, είναι από το Ιράκ και μεταξύ και γύρω στις 8.000 από άλλες χώρες, εκ των οποίων έχουμε και καμιά τρακοσαριά από ξένους μαχητές, παιδιά ξένων μαχητών Ευρωπαίων. 300 Γάλλοι, μόνο για τη βορειοανατολική Συρία, 200 από την Ολλανδία, 160 από το Βέλγιο, 60 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γερμανία, Σουηδία, σημαντικούς αριθμούς κρατουμένων. Αλλά δεν έχουμε δει ε, πόσα παιδιά. Δεν έχουμε δει στοιχεία. Είναι στην καταβλήμα σε διαφορετική τοποθεσία από ό,τι ενήλικη. 250 αγόρια 9 χρονών ε, κρατούνται μαζί με ενήλικες. Μάλλον όμως τα νούμερα είναι υψηλότερα. Κανένας ε, δεν ε, διώκεται ποινικά και δεν υπάρχει κάποια προοπτική προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τα παιδιά αυτά είναι ευάλωτα. Χρειάζονται κατεπηγόντως προστασία για να μην τους συμβεί περαιτέρω κακό. Πριν την έναξη στρατιωτική επέμβαση, ε, ήδη έλεγε η Εξεταστική Επιτροπή ότι υπάρχει τραγική κατάσταση εκεί. Και σίγουρα μετά τι αρχέ Οκτωβρίου τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι κίνδυνοι για την προσωπική ασφάλεια των παιδιών, ε, για δημιουργία ψυχολογικών τραυμάτων και από πήρε στρατολόγησης και κακοποίηση του. Ήθελα να σας τα πω όλα αυτά για να σας δείξω ότι βλέπουμε τι ζουν άλλες χώρες, αλλά και να σας πενθυμίσω ότι είναι αναγκαίο να επαναπατριστούν οι ξένοι και οι οικογένειές της. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό. Οι περισσότεροι ξένοι Ιρακινοί είναι από Ιράκ, Βόρεια Αφρική, Κάφκασο και άλλες περιοχές. Και πολύ συχνά γενική συζήτηση για το θέμα αυτό λέει ότι οι χώρες της Ένωσης αστικά φέρνουν το μεγαλύτερο βάρος, όμως δεν θα πρέπει ε, τη συζήτηση να την ε, στρέφουμε σε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά να βλέπουν ποια είναι τα προβλήματα και τι λύσεις μπορούν να δοθούν για να λυθεί το ανθρωπιστικό πρόβλημα. Η πρωταρχική ευθύνη λοιπόν είναι, σύμφωνα και με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, να ληφθεί υπόψη το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Αυτό σημαίνει επαναπατρισμό Άρα θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα κράτη τις προσπάθειές τους για να παράσχουν προξενική συνδρομή ε, και αν χρειαστεί να βοηθήσουν να καθοριστεί η θαγήνα των παιδιών και να ε, διευκολύνουν την αξιοπρεπή ε, επιστροφή των παιδιών στις χώρες καταγωγής τους, τον απατραπατισμό τους. Πρέπει να κυριαρχεί η αρχή της οικογενικής επανένωσης και μη επαναπρόθεσης για τα παιδιά. 17 χώρες τουλάχιστον ήδη έχουν επαναπατρίσει πάνω από 600 650 ε, παιδιά που ζουν μαζί με συγγενείς τους, κυρίως με τις μητέρες τους που επέστρεψαν ε, στην Ένωση. Θα μπορούσα να μην είναι ακριβή βέβαια τα στοιχεία αυτά, γιατί δεν τα έχω ακριβώς. 8 ε, με 9 χώρες, πολύ λίγα παιδιά έχουν επαναπατρίσει μέχρι τώρα συνολικά. Ενώ σε σύγκριση με το μέγεθος του πληθυσμού των υπηκών των χωρών του ε, στου καταβλισμού, στα στρατόπεδα. Αυτό γίνεται συνήθω κατά περίπτωση και πρόκειται κυρίω για συνόδευτα παιδιά. Τα νεότερα συνήθω, τα πιο μικρά, που δεν φαίνεται να έχουν εμπλακεί ε, σε τέτοιου είδου δραστηριότητε που ε, σχετίζουν του ξένου μαχητέ. Η σχέση λοιπόν μεταξύ ενός ε, θύματος και ενός φερόμενου ως δράστη είναι δύσκολο ε, για τα παιδιά. Μπορεί να είναι θύματα κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, μπορεί και κάποια να έχουν κάνει κάποια αξιόπινη πράξη. Είναι όμως παιδιά κάτω των 18 και πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίζονται ως θύματα. Τα παιδιά που πάνε σε τρομοκρατικέ ομάδες ζουν υποδεινή κατάσταση, εξαναγκάζονται, εκφοβίζονται. Ε, είναι θέμα επιβίωσής τους. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι, τα κίνητρα για την συμμετοχή τους σε τέτοιες ομάδες. Χρειάζεται ατομική αξιολόγηση και διαλογή για αυτούς τους νέους. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση και στην επανένταξη Φαίνεται ότι η αρχική διαλογή γίνεται από τι συριακές δημοκρατικές δυνάμεις σε κάποιους καταβλισμούς. Δεν συνάδουν όμως με τα διεθνή πρότυπα και οι αρχές αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες να ελέγξουν τα στρατόπεδα και τους καταβλισμούς αυτούς. Η τουρκική ε, επιχείρηση σίγουρα ε, δημιούργησε πολύ μεγαλύτερες πιέσεις Πολλές χώρες ε, διαπραγματεύονται με το Ιράκ ε, την ε, επιστροφή των υπηκών τους να δικαστούν εκεί ή στην περιοχή. Αυτό όμως δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες ότι δεν θα είναι δικές οι δίκες και θα οδηγήσουν σε θανατικές καταδίκες και αυτό αντιβαίνει στα πρότυπα του ΟΗΕ και στο διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση. Δεν μπορεί ε, να παραμένει η Δύση αδρανής. Πρέπει να γίνεται λοιπόν ε, η σωστή διαλογή και αξιολόγηση και να υπάρχει κοινωνικο-οικονομική φροντίδα για την απανένταξη αυτών των ατόμων. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πρόσβαση σε ένδικα μέσα, αποκατάσταση, επανένταξη, όλα αυτά μπορεί να τα εξασφαλίσει μόνο η Δύση και έτσι θα ελαφρύνει την τραγική κατάσταση επιτόπου. Σας παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος, να ολοκληρώνετε σιγά σιγά, κυρία Παρά. Ωραία, τότε να ολοκληρώσω λέγοντας τα εξής. Να δούμε ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Η επιτακτική ανάγκη αποτροπής η πρόεδρος τρομοκρατίας. Ο Υπουργό ε, Οικονομικών ε, της Ολλανδίας είπε ότι οι ξένοι μαχητές ε, είναι ξένοι μόνο για τη χώρα στην οποία ταξιδέψαν, αλλά είναι συμπατριώτες μας, είναι γνωστοί μας, σύντροφοι, μάλλον συμμαθές των παιδιών μας παιδιά που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, ανήκουν στις κοινωνίες μας. Αυτό είπε. Επομένως, το να μην επαναπατριστούν παρά την πάρα πολύ κακή κατάσταση επιτόπου θα πυροδοτήσει περαιτέρω κινητοποίηση τέτοιων ξένων μαχητών. Και θα στιγματίσει πολύ κόσμο. Ε, ήδη ε, πρέπει να σας πω ότι και στα στρατόπεδα γίνεται ισοσπαστικοποίηση των παιδιών, άρα δεν πρέπει να παρατείνουμε την οδύνη των παιδιών, την έκθεσή τους ε, στην ε, τρομοκρατική διδαχή. Και Επίσης σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως η στρατιωτική επέμβαση κατέστη ε, προβληματική την ασφάλεια στα στρατόπεδα ε, κράτησης. Πολλοί έχουν τραπετεύσει από τους ξένους μαχητές. Μπορεί κάποιοι να ανησυχούν για το τι θα γίνει ε, πίσω στις χώρες αν τους επαναπατρίσουν. Μήπως όμως ο μη επαναπατρισμός τελικά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα γιατί δραπετεύουν πολλοί ξένοι μαχητές ε, και επίσης ε, υπάρχει κίνδυνος ε, να στρατολογηθούν και νέα παιδιά και να δημιουργηθεί μια νέα γενιά τρομοκρατών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ οι εγγεγραμμένοι. Εάν ο καθένας ξεπερνάει τόσο πολύ το χρόνο του, δεν θα μπορέσουν κάποιοι καθόλου να πάρουν το λόγο. Γι' αυτό σας παρακαλώ όλους, τονίζω όλους, να μην ξεπερνάνε το χρόνο σας. Δέκα λεπτά έχουμε δώσει ε, για τον κάθε εισηγητή. Στα δέκα λεπτά θα, θα κόψω το μικρόφωνο. Η κυρία Κριστιαν Χοέν είναι Principal Advisor ε, και συν, στο συντονιστικό όργανο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ Μαϊτέ. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική για τον επαναπατρισμό των ε, ε, τρομοκρατών και των παιδιών των τρομοκρατών στο Συρία και το Ιράκ. Πρόκειται για ένα θέμα εθνική ασφάλεια, το οποίο τα κράτη-μέλη θέλουν να το αποφασίζουν τα ίδια. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό για τα κράτη-μέλη, λοιπόν. Τα κράτη-μέλη έχουν επαναπατρίσει παιδιά από στρατόπεδα από τη Συρία και το Ιράκ. Κατά περίπτωση εξέτασαν όμω. Και κυρίω πρόκειται για συνόδευτου ανηλίκου. Και κάποιες γυναίκες επίσης επαναπατρίστηκαν. Χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μία ομάδα 7 κρατών εξετάζει τι γίνεται στην περιοχή και εξετάζει τη δημιουργία ενός άνω του δικαστηρίου με το Ιράκ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δραστηριοποιηθεί σε ό,τι αφορά τη Συρία και το Ιράκ και την επατρεπατισμό των ε, μελών. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά να σας πω ποιες είναι οι συνέπειες της ε, απόφασης του Πρόεδρου Τραμπ και να δούμε μετά τι γίνεται και στα στρατόπεδα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο λοιπόν ε, ευαισθητοποίηση για την ε, ριζοσπαδικοποίηση, έχει προτείνει κάποιε καλέ πρακτικέ για το πώ θα αντιμετωπίσουμε του αλλοδαπού μαχητέ και τι οικογένειέ του που είναι αναπατρίζονται. Και υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για τα παιδιά σε ό,τι αφορά και την ψυχολογική αντιμετώπιση τους. Κάποια παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει από εμπόλεμες ζώνες. Κάποια κρατημέλη όπως η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν και κάποιες ιδιαίτερες υπηρεσίες που υποδέχονται τα παιδιά αυτά και συνοδεύουν την επαρένταξή τους. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ δίνει ανθρωπιστική βοήθεια στα, στους καταβλισμούς στη Συρία και παρά το κουρδικό μέτωπο συνεχίζει η, συνεχίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια με το ντόπιο προσωπικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, προσπαθεί να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για την ασφάλεια των συνόρων, για τις έρευνες, για την εισαγγελία. Μία από τις προκλήσεις στην επαναπατρισμό είναι να πιστούν οι γυναίκες και ε, τα μέλη των οικογενειών σε ό,τι αφορά τις ποινές. Ε, στη Γενική Διεύθυνση Home έχει διοργανωθεί ένα εργαστήριο τον Ιούλιο μαζί με τις ΕΠΑ και συλλέξαμε πολλές πληροφορίες και η Europol επίσης έκανε μια πρώτη, δημιούργησε μια πρώτη μονάδα κρούσης για τον επαναπατρισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει βοήθεια και σε χώρες όπως την Ισία σε ό,τι αφορά την υποδοχή ξένων μαχητών και των οικογενειών τους και επίσης ε, διοργανώθηκε ένα σεμινάριο για να κοιτάξουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, δώσει μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερη υποστηρίξη. Και επίση, ε, μία από τι προσπάθειε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει πιο συνεκτικές πληροφορίε σε ό,τι αφορά και την Ιντερπολ για τους φυλακισμένους ε, στην Ιορδανία σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της Ιντερπολ για τους, τα σύνορα και στα Δυτικά ε, Βαλκάνια επίσης για τις κινητές συσκευέ. Όλα αυτά λοιπόν παρέχουν υποστήριξη πέρα από την ιδεολογική συζήτηση σε ό,τι αφορά την ε, τους αλλοδαπούς μαχητές μία θαλάσσια άσκηση της Interpol ε, ε, ανακάλυψε πάνω από δεκάδες μάλλον ε, μετανάστες αλλοδαπούς μαχητές οι οποίοι ταξίδευαν στην Μεσόγειο. Κατά δεύτερον, τι σημαίνει η απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να αποσύρει τα στρατεύματα από τη Συρία, η δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης, η συμφωνία μεταξύ του κουρδικού SDF και του Νασάντ υπό τη ρωσική αιγίδα έχει δημιουργήσει νέους όρους και νέες συνθήκες. Και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέα ορισμό πολιτικής. Πολλά στρατόπεδα είναι υπό το STF στην παρούσα Η ανθρωπιστική κατάσταση στα στρατόπεδα φαίνεται ότι έχει ήδη δυσκολέψει παραπάνω. Υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια. Καταρχάς, να ξεφύγουν από τη φυλακή, να αποτράσουν οι αλλοδοποί μαχητέ. Και τα γυναικόπαιδα. οι αρχέ των ΗΠΑ δήλωσαν ότι περίπου 100 αλλοδοποί μαχητέ ήδη έχουν τραπετεύσει από τι φυλακέ στη Συρία και επίση 800 περίπου γυναικόπαιδα έχουν ε, φύγει. Οι αλλοδοποί μαχητέ έχουν ε, συλληφθεί από την Τουρκία και έχουν ε, επιστραφεί στις ε, χώρες τους ενδεχομένω φυσικά και ο Ασάντ να χρησιμοποιήσει τους αλλοδαπούς μαχητές ως ε, νόμισμα για ανταλλαγή ή και να το εκτελέσει. Είναι σημαντικό οι αλλοδαποί μαχητέ και οι οικογένειέ του να εντοπίζονται στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συντονιστή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλαν επιστολή για να υπάρχει καλύτερη ροή πληροφοριών στο σύστημα Σέγγεν, το οποίο λαμβάνουν από τη ΣΥΠΑ μείωση τη Ιντερπολ και σε ό,τι αφορά του αλλοδαπού μαχητέ που δεν είναι Ευρωπαίοι. Και καλούμε λοιπόν τη ΣΥΠΑ να μοιράζονται πληροφορίε μαζί μα. Έχουμε ένα σύντομο χρονικό περιθώριο κάποιων μηνών όσο οι αλλοδαποί μαχητέ και οι οικογένειε του είναι υπό τον έλεγχο του STF. Να το χρησιμοποιήσουμε προκειμένου η ΕΚΟ, για παράδειγμα, να δώσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι, η πρόεδρος διακόπτη, Μήπω θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί σα παρακολουθούν οι διερμηνεί. Η ΕΚΟ λοιπόν θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στα στρατόπεδα και ίσω όταν δυνατόν να γίνονται και μελέτε, ε, ε, μάλλον αξιολόγηση κινδύνου για τι οικογένειε που είναι μέσα στα στρατόπεδα και να υπάρχουν και κάποια προγράμματα ήδη απασχόληση, ήδη να διαχωριστούν κάποιε γυναίκε οι οποίε ενδεχομένω να θέλουν να ενταχθούν από τι πιο ριζοσπαστικοποιημένε, οι οποίε ασκούν πίεση στι άλλε. Κάποιε γυναίκε είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικοποιημένε και. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά τώρα, τα παιδιά στα στρατόπεδα στη Συρία, συχνά είναι πάρα πολύ μικρά σε ηλικία. Πολλά και κάτω των 6 ετών. Και τα παιδιά είναι κατά πρώτον θύματα. Κάποια έχουν ήδη διαποτιστεί από τις ιδέες ε, που τους δίνουν οι μητέρα τους σε ό,τι αφορά για παράδειγμα Οι γυναίκε λοιπόν είναι αυτές που πολλές φορές χρησιμοποιούν στις συμμορίες του χαλιφάτου τα παιδιά. Οι ψυχολόγοι διατείνονται ότι όσο πιο νεαρά είναι τα παιδιά τα οποία επαναπατραγίζονται, τόσο το καλύτερο, τόσο πιο εύκολο, τόσο πιο πιθανόν είναι να μπορέσουν αυτά τα παιδιά που έχουν υποστεί μεγάλο τραύμα να ενταχθούν στην κοινωνία. Όσο πιο μεγάλα είναι σε ηλικία, τόσο πιο μεγάλο είναι ο κίνδυνο επαναπατρισμού, ε, συγγνώμη, ριζοσπαθικοποίηση και είναι λιγότερο πιθανή η ένταξή τους. Άρα, από πλευρά ασφάλεια καλό θα ήταν να επιστραφούν τα παιδιά αυτά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπάρχουν κάποιε δικαστικέ αποφάσει σε κάποιε χώρε που υποχρεώνουν τι κυβερνήσει, να κάνουν ό,τι μπορούν να επαναπατρίσουν τα παιδιά και τι μητέρες του σε κάποιε κάποιες περιπτώσεις. Το θέμα όμω αυτό είναι περίπλοκο. Υπάρχουν τρει προκλήσει. Η πρώτη είναι ότι πολλοί διαθέτονται ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τα χωρίσουν από τι μητέρε του. Ωστόσο, οι μητέρε του συχνά είναι πολύ ακραίε ριζοσπαστικοποιημένε. Είναι δύσκολο λοιπόν επίση σε πολλέ περιπτώσει να εντοπιστεί η ριζοσπαστικοποίηση. Υπάρχει ένα δισταγμό λοιπόν από τα κράτη-μέλη να επαναπατριστούν και οι μητέρε μαζί με τα παιδιά. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν το βασικό θέμα. Ποια είναι το καλύτερο συμφέρον, το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, να μείνει με τη μητέρα ή να επιστραφεί στην Ευρώπη και να ζήσει με άλλα μέλη της οικογένειάς του. Η δεύτερη πρόκληση είναι η εξή. τώρα το STF δεν έχει επιτρέψει επαναπατρισμό των παιδιών χωρίς τι μητέρες του. Και ω εκ τούτου. Και για το λόγο λοιπόν αυτό τα κράτη-μέλη έχουν το θέμα αυτό των επαναπατρισμού των ασυνόδευτων ανηλίκων. Τρίτη πρόκληση. Χωρίς με αμερικανικά στρατεύματα επιτόπου, πώ θα μπορούσαμε πρακτικά να το οργανώσουμε το θέμα της, ε, του επαναπατρισμού των παιδιών. Όσο υπάρχει αυτό το παράθυρο πριν ε, την ανάληψη του θέματος από τον Ασάντ. Μία γυναίκα η οποία έφυγε με ένα δίχρονο παιδί από στρατόπεδο SDF, πήγε στα σύνορα στην Τουρκία και εκεί βοηθήθηκε από τις ε, ειδικές δυνάμεις τη Ιρλανδίας για να επιστρέψει στην Ιρλανδία και να επαναπατριστεί το παιδί όλος ιδιαίτερος. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά των Αλδαπών μαχητών στη Συρία και στο Ιράκ είναι πολύ περίπλοκα. Από πλευρά ασφάλεια, καλύτερα ήταν, θα ήταν να επιστραφεί και να επαναπατριστεί γρήγορα το παιδί. Αλλά δεν είναι απλό και η απόφαση του STF να απαγορέψει την επαναπατρισμό των παιδιών χωρίς τις μητέρες του, περιπλέκει τα πράγματα. Και προφανώς ανησυχούμε κι εμείς για τη μοίρα των παιδιών αυτών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χοένα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πολ Βαν Τίχελτ, ο οποίος είναι διευθυντής της συντονιστικής μονάδας για την ανάλυση της απειλής, την ΟΚΑΜ του Βελγίου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την ε, την πρόσκληση που μου απευθύνεται. Ε, δεν θα ξεπεράσω τα 10 λεπτά, ελπίζω, γιατί νομίζω ότι είχα ήδη την ευκαιρία να εκφράσω την ε, βελγική άποψη για το θέμα αυτό ήδη το 2018. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι μια ερώτηση προς όλους. Πόσο θα συνεχίσουμε, ε, ε, για πόσο ακόμα θα συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Εδώ και κάποια χρόνια ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ε, πότε θα σταματήσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και άλλωστε τα έχουμε πει όλα όσον αφορά αυτά τα ευαίσθητα ανθρωπιστικά ζητήματα. Εγώ είμαι διευθυντής τη συντονιστική Μονάδα για την ανάλυση της απειλή ε, και δουλειά μου είναι να μαζεύω όλες τις πληροφορίες ε, και να αξιολογώ ε, την απειλή καθώς επίσης ε, και να υποβάλω προτάσεις ε, για ε, τις στρατηγικές εξελίξεις και για τις στρατηγικές προτάσεις. Αυτή είναι η δουλειά μου και φαντάζομαι ότι γι' αυτό με καλέσατε εδώ. Κύρια δουλειά μου λοιπόν είναι να διευκολύνω τον συντονισμό όλων αυτών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που απορρέουν από την ριζοσπαστικοποίηση. Δεύτερο, ε, η αξιολόγηση της ε, ε, απειλής είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τους ξένους μαχητές, αλλά η μεγαλύτερη απειλή για, τους, για την Ευρώπη προέρχεται στην ουσία από τους ε, λεγόμενους μοναχικούς ε, λύκους, ε, αυτούς δηλαδή τους μεμονωμένους ανθρώπους οι οποίοι εμπνεόμενοι από τα όσα συμβαίνουν στις χώρες που μας απασχολούν ξεκινούν να κάνουν κάποιες δικές τους δράσεις. Τρίτον, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το λάθος να βάλουμε όλους σε ένα ίδιο καλάθι. Ε, εμένα δικιά μου δουλειά είναι να βλέπω αντικειμενικά ε, και να αναλύω αν, ε, αντικειμενικά τις καταστάσεις ανεξάρτητα από το πόσο έχουν τραυματιστεί οι χώρες όπως ας πούμε το Βέλγιο την 22 Μαρτίου του 2016 γιατί πολλές φορές ε, οδηγός μας στις συζητήσεις ε, είναι αυτή η συναισθηματική, ας πούμε, η συγκινησιακή ε, σκέψη. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ε, αντικειμενικοί επίσης, ε, να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Ένα παιδί δύο ετών δεν είναι το ίδιο με ένα νέο 16 ετών. υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν τραυματιστεί από την σκληρότητα και την ομότητα που έχουν δει γύρω τους, άλλα όμως που έχουν ε, ζήσει ναι, την ε, κατάσταση αυτή. Ε, από όσο ξέρουμε εμείς, τα περισσότερα παιδιά είναι 2, 3, 4 ετών ε, και θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια μικρά παιδιά δεν είναι ένα πρόβλημα ασφάλειας, είναι ένα πρόβλημα ανθρωπιστικό. Ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα το οποίο ε, ήδη προϋπήρχε της ε, νέας κατάστασης, ε, αυτή που προέκυψε δηλαδή πριν μερικές εβδομάδες, με την απόρριση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την Συρία. Ε, εδώ και μήνες, για να μην πω εδώ και χρόνια, τα κέντρα μας λαμβάνουν πληροφορίες ε, και μέσω ιδιωτικών ιατρικών βελγικών αποστολών ε, λαμβάνουμε, λέω, στοιχεία και καταγγελίες για παιδιά τα οποία ζουν σε κατάσταση υποσυτισμού ή πολύ κακών συνθηκών διατροφής, παιδιά τα οποία προσπαθούν να τα προσιλητήσουν διαρκώς οι μητέρες τους ε, οι οποίες ε, είναι άκρως ριζοσπαστικοποιημένες, αλλά αυτό αναφέρθηκε ήδη. Πιστεύω ότι μέσα από το πρίσμα της προληπτικής κοινωνικής αντιμετώπισης θα πρέπει να προσεγγίσουμε ε, τα παιδιά αυτά. Τον Ιούνιο αυτού του έτους είχαμε κάποιους επαναπατρισμούς και στο Βέλγιο ε, έχουμε το μεγάλο, η μεγάλη πολυτέλεια, όπως και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να είμαστε ε, αρκετά πλούσιες χώρες, που σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε κοινωνική πρόνοια στα παιδιά αυτά. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Πραγματικά μέσα και από τις υφιστάμενες δομές των δικαστηρίων των νέων και άλλων παραπλήσιων δομών και στη ε, και στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο Βέλγιο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των παιδιών αυτών. Βεβαίως, όπως υπόθηκε και προηγουμένως ε, και από την Κριστιαν, ε, υπάρχουν διαφορετικές σκοπιές. Υπάρχει βεβαίως η σκοπιά της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης των παιδιών, αλλά υπάρχουν πολιτικά, γεωπολιτικά ζητήματα και άλλου είδου θεωρήσει γιατί δεν πρέπει να μιλήσουμε μόνο για τα παιδιά, μιλάμε και για τις μητέρες και για τους ε, πατεράδες ε, και εκεί η κατάσταση είναι διαφορετική και σε αυτούς, ε, για την περίπτωση αυτών των γονιών δηλαδή, η πολιτική συνένεση είναι σαφώς μικρότερη. Όπως είπε και στην αρχή, θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ξεχωριστά το καθένα και να μην βάζουμε στο ίδιο καλάθι τους πάντες και τα πάντα. Και όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο τρόπο για τους Βέλγους ε, και Ολλανδούς συναδέλφους. Ε, όσον αφορά αυτούς που βρίσκονται ήδη εδώ και δύο χρόνια, μητέρες που βρίσκονται σε στρατόπεδα ε, εδώ και δύο χρόνια, έχουμε ε, πληροφορίες ότι αυτές έχουν αποκηρύξει την ιδεολογία, αυτές που βρίσκονται δηλαδή στα στρατόπεδα αυτά πάνω από δύο χρόνια. αλλά βεβαίως είναι γεγονός ότι έχουμε και άλλες πληροφορίες, ότι ενδεχομένως στα στρατόπεδα αυτά και μεταξύ και αυτών των γυναικών μπορεί να υπάρχουν ακόμα σκληροπυρηνικές ριζοσπαστικοποιημένες γυναίκες. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα, μία ακόμα παρατήρηση. Γιατί νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε ήδη ε, μία παρατήρηση από τη βελγική ας πούμε σκοπιά, μία χώρα, το Βέλγιο, μια ακομα παρατηρηση γιατι νομιζω οτι δεν αναφερθηκε ηδη μια παρατηρηση απο χώρα που βρίσκεται στο κέντρο ε, της Ευρώπης. Κατά τη δική μας άποψη, αυτά τα δύσκολα και ευαίσθητα θέματα απεικονίζουν στην ουσία την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας. Όχι συνεργασία μονάχα σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί υπάρχει ανάγκη για ε, κοινή ε, αν όχι ευρωπαϊκή, τουλάχιστον πολυμερή προσέγγιση αυτών των ιδιαίτερα ευαίσθητων θεμάτων. Ε, τα έχουμε πει, αλλά θέλω να το ξαναπώ κυρίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο τελικά να έχουμε ε, τις τελευταίες εβδομάδε ε, μετά τα ε, γεγονότα τα τελευταία. Έχουμε μεγάλη δυσκολία να βρούμε ασφαλείς αξιόπιστες πληροφορίες. Επομένως είναι σημαντικό να είμαστε συντονισμένοι και όσον αφορά και τα όσα κάνουμε με τη Συρία, με το Ιράκ, με τη ε, Τουρκία. Θα πρέπει να υπάρξουν συστήματα επαναπατρισμού. Είναι πολλές χώρες ε, οι οποίες έχουν επαναπατρίσει ε, παιδιά. Αναφέρθηκε και προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ δύσκολες, ιδιαίτερα ευαίσθητες αυτές οι διαδικασίες επαναπατρισμού και νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί δεν ξέρουμε αρκετά. Διεθνή συνεργασία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί ε, μάθαμε ότι όσο μεγαλύτερη ε, ανταλλαγή πληροφοριών έχουμε ε, για τους ξένους μαχητές μέσω της Interpol, της Europol, των δικών μας εθνικών συστημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια αυτά να έχουμε βιομετρικά χαρακτηριστικά, γιατί οπωσδήποτε στην επιχειρησιακή ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Εμείς από τη ιατρική πλευρά έχουμε ήδη ε, βελτιώσει, μερικές φορές μάλιστα με θεαματικό τρόπο αυτή τη συνεργασία, αλλά ωστόσο θα πρέπει να επαγρυπνούμε και θα πρέπει να είμαστε διαρκώς επικριτικά κείμενοι απέναντι στους εαυτούς μας και να αναρωτιόμαστε διαρκώς ε, αν ε, κάνουμε κάτι σωστά και αν κάνουμε κάτι όπως πρέπει. Το θέμα είναι ότι τούτο το ζήτημα σαφώς ε, μπορεί να είναι περίπλοκο. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα παιδί από Βέλγο πατέρα και Ολλανδή μητέρα και μετά ο Βέλγος πατέρας έχει πεθάνει, ε, ε, η οικογένεια έχει διευρυνθεί με κάποια γαλλικά μέλη και καταλαβαίνετε γιατί λέμε ότι θα πρέπει να τύχει ευρωπαϊκής προσεγγίσεως το θέμα αυτό. Αυτά και στη διάθεσή σας είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συμμεριζόμαστε τα όσα λέτε. Ε, πιστεύουμε ότι ναι, πρέπει να δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα, θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ζακλίν Χάλ, η οποία είναι επικεφαλής ε, της ε, Ένωσης Save the Children. Παρακαλώ. Thank you very Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω την ε, οπτική γωνία μια ε, λειτουργική ε, ΜΚΟ που λειτουργεί στην Συρία για να δώσει κατεπίγουσα βοήθεια στα παιδιά. Το... Η οργάνωσή μας επέτρεψε σε πολλά παιδιά να φτάσουν σε... να πάρουν βοήθεια στην βορειοανατολική Συρία Εργαζόμαστε με χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κλιμάκωση. και αυτό λόγω της σύνδεση και με εμπόλεμε οργανώσει όπω η ISIS. Θα ήθελα να παρουσιάσω πώς έχει κατάσταση και να πω μετά τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Έχουμε σήμερα 12.300 αλλοδαπούς μη Σύριους και μη Ρακινούς ε, στη βορειοανατολική Συρία. 9.000 περίπου παιδιά από 40 εθνικότητες από κάθε περιοχή στον κόσμο. Οι, τα παιδιά αποτελούν το βασικό καθήκον μας ε, και πάνω από 4.000 ε, παιδιά είναι κάτω από την ηλικία των 5. Η κλιμακούμενη Λιβύα στην Συρία έχει επιθυνώσει περαιτέρω την κατάσταση των παιδιών αυτών στιγματισμένα είναι, είναι σε μία διάμεση κατάσταση για την ενσωμάτωσή τους. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους ε, είναι σε δύο στρατόπεδα, αλχόλ και ουόρς. Στο αλχόλ. 68.000 άτομα ζουν εκεί. Οι αλλοδαπές ε, οικογένειες ε, έχουν λάβει έχουν βοήθεια από την ISIS σε ό,τι αφορά άτομα τα οποία έχουν ζήσει υπό την προστασία του ISIS. Το Save the Children είναι η μοναδική μοικείο εκεί. Παρέχουμε εκπαίδευση, διατροφή, τρόφιμα και διαχείριση των παιδιών. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο κόσμος έχει περιορισμένη πρόσβαση σε σωστή τροφή. Δεν υπάρχουν ε, παρκή καταλήμματα. Ο κόσμος παρακαλά να έχει μια σκηνή και είναι περιορισμένη και η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ε, υγιεινής. Επίσης, περιορισμένη ε, πρόσβαση έχουν τα παιδιά ε, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Είναι φτωχέ οι συνθήκε υγιεινή. Αυτό οδηγεί σε κίνδυνο ξεσπάσματο μολυποθικών ασθενειών. Έχουμε επίση μεγάλε ελλείψει σε βιταμίνε. Τα παιδιά δεν έχουν ασβέστη λόγω έλλειψη γάλακτος και γαλακτοκομικών, τα παιδιά ε, τους πέφτουν τα τόντια και είναι σε τραγική κατάσταση. Μία νεαρή μητέρα, η οποία μεταφέρθηκε από τους γονείς της ως παιδί στην Συρία, ε, είδε τον πατέρα της να αποκεφαλίζεται από την Άισις και στη συνέχεια την ε, έβαλε το ISIS να παντρευτεί καταναγκαστικά και να μείνει αγκίωσα. Θέλω μια φυσιολογική ζωή, δεν θέλω άλλη Δεν ε, νομίζω ότι υπάρχει τίποτε πιο όμορφο από αυτό. Το βασικό λοιπόν θέμα εδώ είναι το εξή, ότι τα παιδιά, τα λαταπά παιδιά που είναι στη Συρία απαγιδευμένα είναι θύματα, αθώα θύματα. Ω τέτοια θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουν ε, περάσει από άθλιες συνθήκες και χρειάζονται ειδική βοήθεια για να μπορέσουν να επαναληφθούν σε ένα καθεστώς φυσιολογικότητας, το οποίο είναι δυνατόν να γίνει σε ένα καταβλισμό μεταναστών, προσφύγων, σε μια εμπόλυμη ζώνη. Δεδομένων λοιπόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά, η Save the Children ζητά από, την, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά να επιστρέψουν στις χώρες τους. Πρόσφατα ασκείται μεγαλύτερη πολιτική πίεση σε κρατημέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο για να κάνουν επαναπατρισμό. Για τα παιδιά, υπό το διεθνές δίκαιο, υπάρχει υποχρέωση για τις ε, προξενικές αρχές για τον επαναπατρισμό. Η μη υποβοήθηση λοιπόν του επαναπατρισμού από τις βελγικές αρχές για παράδειγμα, ουσιαστικά σημαίνει ότι αρνούνται στα παιδιά αυτά τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει να καλέσουμε λοιπόν τα παιδιά αυτά να πάνε πατριστούν με τις μητέρες τους, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο πολλά. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπαν πολλοί, έγινε ε, παναπατρισμός ε, παιδιών που αποτελεί και την καλύτερη δυνατή λύση. Αποτελεί νομική και ηθική ευθύνη αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, αναφέρουν και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 24 και το, Σύμβαση για τα Παιδιά ορίζουν όλα ότι είναι απαραίτητο ο επαναπατρισμό. Θα πρέπει λοιπόν τα κρατημέλη να κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να διευκολύνουν τον επαναπατρισμό. Ταξιδιωτικά έγγραφα. Βοήθεια για τη μετάβαση στα σύνορα. Και μεταφορά στα σπίτια του καθενό. Τα κράτη-μέλη μπορούν να δώσουν ένα τέλο στο έλεος, στο, στις συνθήκες αυτές που ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Κάποια κράτη-μέλη ζητούν από τα παιδιά και από τις μητέρες τους να πάνε στα προξενία στο Ιράκ για να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό είναι αδύνατον. Δεν μπορούν να μετακινηθούν. Δεν έχουν την ελευθερία. Ενώ οι αρχές των κρατών μελών έχουν πρόσβαση στα στρατόπεδα των προσφύγων. Ο επανεπατρισμός λοιπόν είναι δυνατός. Αρκεί να υπάρχει πρωτοβουλία των αρχών. Ο επίσης έχει συζητηθεί με το Δημοκρατικό Κουρδικό Συμβούλιο και ο επαναπατρισμός από την βορειοανατολική Συρία είναι ακόμα δυνατός. Τα δύο στρατόπεδα λοιπόν είναι εκτός της εμπόλεμης ζώνης, είναι υπό κουρδικών αρχών, υπό κουρδικής αρχής και υπάρχει πρόσβαση. Είναι ασφαλές το στρατόπεδο και αυτό θα πρέπει να το εξετάζουμε φυσικά κάθε μέρα. Είναι ανοιχτά τα σύνορα προς το Ιράκ, υπό κουρδικό έλεγχο. Αν και αυτό μπορεί να αλλάξει αν αναλάβει τον έλεγχο η κυβέρνηση της Συρίας. Έχουμε και ένα τρίτο στρατόπεδο στην Ίσα, όπου Έφυγαν όμως από εκεί οι οικογένειες γιατί επικράτησε σύγχυση. Εκατοντάδες λοιπόν γυναίκες και παιδιά έχουν φύγει από τον καταβλισμό αυτό και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Γι' αυτό θα πρέπει ο επαναπατρισμός να λάβει χώρα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο κάλεσε πρόσφατα τα κράτη-μέλη και παραθέτω να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση και στις ανάγκες των Ευρωπαίων παιδιών που έχουν γονείς ε, μαχητές ISIS προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα βασικά δικαιώματά του και να έχουμε κατά νου το συμφέρον των παιδιών σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί για τα παιδιά. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ποτέ δεν είναι προς το συμφέρον ενός πεντάχρονου παιδιού να μένει σε ένα στρατόπεδο προσφύγων χωρίς να έχει καμία πρόσβαση σε φαγητό, σε εγκαταστάσεις οικονομικής περιθαλψής και ο χάρτης των θεμελιδών δικαιωμάτων ορίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υλοποιήσει το ψήφισμα του για την επιστροφή των παιδιών αυτών στην χώρα προέλευσης. Θέλουμε λοιπόν ηγεσία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα σαφές μήνυμα προς τις κυβερνήσεις να δράσουν τώρα πρώτα τα πράγματα πάνω στο προχώρητο. Τέλος, σε ό,τι αφορά την επιστροφή των παιδιών χωρίς τις μητέρε του. Ω συμβαστική λύση σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει λόγος η πολιτική του επαναπατρισμού να περιοριστεί σε ασυνόδευτα παιδιά. Ούτε να επιβάλλεται μια διαδικασία εξέταση κατά περίπτωση που παίρνει χρόνο Όλα τα παιδιά θα πρέπει να επιστραφούν. Τα παιδιά με τις μητέρες τους είναι εξίσου αθώα με όλα τα άλλα παιδιά. Οι μητέρες αυτές είναι το μοναδικό σταθερό στοιχείο στη ζωή τους. Δεν ζήτησαν να πάνε στη Συρία, ούτε ζήτησαν να γεννηθούν στη Συρία. Ο επαναπατρισμός είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουν τα παιδιά αυτά για να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Θα πρέπει λοιπόν το συμφέρον των παιδιών να έχουμε κατά Θα πρέπει να κάνουμε το βήμα αυτό προς τον επαναπατρισμό και να προασπιστούμε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τις διάφορες ε, προοπτικές ε, και οπτικές για το θέμα. Έχουμε έναν πάρα πολύ μακροσκελή κατάλογο ομιλητών. Οι συντονιστές θα έχουν στη διάθεσή τους δύο λεπτά έκαστος, οι υπόλοιποι ένα. Και θέλω να σας πενθυμίσω δύο πράγματα. Μιλάμε για παιδιά, πρώτο. Έτσι μην το ξεχνάτε, για αγόρια και κορίτσια. Και δεύτερον, είμαστε σε μια αίθουσα που υπάρχουν συγγενείς ορισμένων από αυτά τα παιδιά. Άρα με, καταλαβαίνετε την οδύνη τους. Θα είμαι πολύ αυστηρή με το χρόνο και με τον κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Ο κύριος Πίτερς έχει το λόγο μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσαν και για τις απόψεις τους. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και πάρα πολύ λεπτή, ευαίσθητη συζήτηση και σημαντικότατη. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είναι απαράδεκτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση νέα παιδιά, μικρά παιδιά, να βρίσκονται σε τόσο δύσκολη κατάσταση σε στρατόπεδα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ένας από τους ομιλητές ε, είπε ήδη ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Και κάποια στιγμή θα εκπνεύσει η προθεσμία. Το παράθυρο, το χρονικό θα κλείσει. Οι αξίες για την Ένωση είναι πολύ σημαντικές, ιδίως όταν μιλάμε για μικρά παιδιά. Δεύτερον, τίθεται το ερώτημα τι αρμοδιότητε έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα θέματα. Ο ε, κύριος ε, Βαντίχελτ μίλησε για την ε, πολυμερή προσέγγιση, λέγοντας ότι ίσω να είναι πιο αποτελεσματική. γιατί η Ένωση δεν έχει τη νομική βάση ή ίσως επαρκείς αρμοδιότητες ως προς αυτό, άρα χρειάζεται μια διεθνής προσέγγιση. Και ποια είναι τα βήματα προς κάτι τέτοιο είναι η ερώτησή μου, αν υιοθετηθεί αυτή η πολυμερής προσέγγιση. Επειδή επίσης έγινε λόγος για ανάγκη ανταλλαγής δεδομένων από τα διάφορα κράτη-μέλη, πώς μπορεί να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό. Και τώρα έχουμε στο τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω. Συγγνώμη κυρία Πέτερς, αλλά δεν έχετε άλλο χρόνο. Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες πρακτικές. Τέλος ο λόγος σας κύριε Πέτερ, συγγνώμη, τι να κάνουμε. Υπάρχει συντονιστή από το Σοσιαλιστές, εσείς, κύριε Μορένο. Μορένο Σάντσεφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε Μαϊτέ. Να ευχαριστήσω και εγώ τους ομιλητές όπως είπες αγαπητή πρόεδρε και το είπε και η Μαρή, πρόκειται κυρίως για παιδιά, πρόκειται για θύματα, ε, για αφρικαλαιότητες ε, που έκαναν οι γονείς τους, αλλά τα ίδια τα παιδιά είναι θύματα και πρέπει να τα προστατεύσουμε. Κύριος Φαντή Χελτή, παιδί πολύ σημαντικά. Πρώτον, χρειάζεται ευρωπαϊκή προσέγγιση, γιατί ναι, κάθε, κάθε κράτος κάνει τα δικά του, αλλά δεν αρκούν αυτά. Και είπατε επίσης πρέπει να σταματήσουμε τα λόγια και να περάσουμε στα έργα και συμφωνώ απόλυτα η Επιτροπή μας και με τις δικές σας τις συμβουλές τι και καθοδήγηση, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα περιμένουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα, να διαθέσουμε τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τον επαναπατρισμό, για την προστασία και την επανένταξη των παιδιών αυτών στην κοινωνία τι να κάνουμε και πώ να το κάνουμε. Σίγουρα εμεί θα κάνουμε πάντα δυνατόν ώστε να συνεργαστούμε και με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να προοδεύσουμε, να προχωρήσουμε μάλλον. Ευχαριστώ σε ευχαριστώ πολύ. Βάλμανς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους διάφορους ομιλητές. Ο κύριος Πάουλ Φαντίνχελτ είπε ότι πριν δύο χρόνια είχαμε ένα στραπαστικό σεμινάριο εδώ για τα δικαιώματα των παιδιών, την κατάσταση των παιδιών σε στρατόπεδα, καταβλισμού, αλλά μιλήσαμε και για την ασφάλεια. Να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για παιδιά σε στρατόπεδα. Τότε στο σεμινάριο πριν δύο χρόνια είχαμε έναν από την Υπηρεσία Πληροφοριών τη Ολλανδίας που μα έλεγε ότι τα μικρή ηλικία παιδιά κάποια από αυτά τους μαθαίνανε ε, να αποκεφαλίζουν την κούκλα τους ε, για να μάθουν να κόβουν κεφάλια. Ε, θα σας σοκάρει αυτό που σας λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν πρέπει να πληρώσουν τα κρίματα των γονέων τους αυτά τα παιδιά, πρέπει να τα πατρίσουμε το στομότερο δυνατόν. Αυτά μου τα λέει η καρδιά μου, αλλά τι μου λέει το μυαλό μου και τι μπορεί να κάνει το Βέλγιο, δεν ξέρω. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα ε, τα οποία θέλω να απευθύνω στον Πάολο Φαντίχελτ από το Βέλγιο, από την Ομάδα Συντονισμού για την Ανάλυση Απειλών. Καταρχά, έχουμε επαρκεί δομέ για να ε, υποδεχθούμε τα παιδιά αυτά, ναι ή όχι. Δεύτερον, έχουμε επαρκεί πληροφορίε για την κατάσταση των παιδιών που ζουν σε αυτά τα στρατόπεδα, αλλά κυρίω για του ξένου ε, μαχητέ ε, που έρχονται από ευρωπαϊκά κράτη. Και τρίτον, μιλήστε για βιομετρικά στοιχεία. Πληροφορίε όμω, ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή δεδομένων υπάρχει μεταξύ των κρατών. Πολύ λίγε πληροφορίες πήρε η Interpol πριν ε, τις επιθέσεις Βρυξέλλες. Και στρέφομαι τώρα σε όλα τα μέλη ε, του πάνελ και όχι μόνο στη μονάδα συντονισμού για την ανάλυση απειλών του Βελγίου. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση, ότι κάποιοι μιλάνε για την ανάγκη προστασίας κοινωνίας κτλ. Το είπε και ο κύριος Πέτερς όμως, ε, εγώ δεν μιλάω για ένα νιωστό ψήφισμα, μία νιωστή τροποποίηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μιλάω για συγκεκριμένε δράσει που αύριο πρέπει να πάρει, ε, να αναλάβει να κάνει ένα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπρικμό, έχει το λόγο. Εκ μέρου των Πρασίνων. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω του ε, ομιλητέ. Ε, είναι πολύ καλή και αναγκαία συζήτηση αυτή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ και εβδομάδε, για να μην πω χρόνια, δεν έχουμε πρόοδο. Σήμερα πράγματι είναι, ο λόγος για, είναι ώρα για έργα. Ε, και όχι για λόγια. Όλοι το υπενθυμίσατε, μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Είπατε πρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είπε ότι πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν οι χώρες για να επαναπατρίσουν τους ξένους μαχητές. Και το Βέλγιο δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει, το λέω ξεκάθαρα. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη και ε, να μην τιμωρηθούν για τα κρίματα των γονέων τα παιδιά. Εμείς ως εκλεγμένοι πρέπει να υπενθυμίζουμε αυτά τα καθήκοντα και πρέπει να κάνουμε τα λόγια πράξης. Είναι και θέμα ασφάλειας, είναι και θέμα πρόληψης. Ο, έλεγξος, ε, το, ο έλεγχος των τραγουδών από τις κουρδικές αρχές δεν είναι εγγυημένος μακροπρόθεσμα. Πρέπει να υπάρχει δικαστική συνδρομή των επαναπατριστέντων. Αυτό το ζητούν όλο και περισσότεροι φορείς και μη εκπροσωπούμενοι σήμερα που προέρχονται από τους δικαστικούς ε, κύκλους τελικά εμπιστευόμαστε ή όχι τα ίδια μας τα δικαστικά συστήματα, γιατί δεν τους επαναπατρίζουμε. Όλοι έχουν δικαίωμα σε δίκαια, αμερόληπτη δίκη μην ε, σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο, τι κάνουμε ε, για να αντιμετωπίσουμε τη βαρβαρότητα. Εμείς έχουμε ευθύνη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Υπάρχουν δυνητικοί τρομοκράτες, ας, πρέπει, το πούμε αυτό, μεταξύ αυτών και υπάρχει κίνδυνος ε, να στρατολογηθούν από το Ισλαμικό κράτος. Και μεταξύ αυτών και τα παιδιά διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο. Πρέπει απέναντι σε αυτή την τρομοκρατία που βλέπουμε εμείς να επανεπιβεβαιώσουμε την πίστη μας στη δημοκρατία. Ευχαριστώ. δεν ξέρω ποιο θα μιλήσει, ο κ. Κόφου, ο κ. Μπέργκ. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Okay. Um, Συνάδελφοι, μετά από την αφέλεια πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Μιλάμε για παιδιά. Παιδιά και άνθρωποι κάτω των 18. Είναι σαφές. Ε, ε, οι μαχητές του ε, ίσης χρησιμοποιούν ακόμα και παιδιά 3-4 ετών για να δολοφονήσουν μειονότητες για τους ομοφιλόφιλους που τους έχουν στο στόχαστρο. Πραγματικά φρικτά πράγματα. Το πρώτο μας καθήκον λοιπόν είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, όχι τους μαχητές των, του ίσης τα παιδιά τους. Θα ήθελα να αναφέρω την έκθεση των Ολλανδικών Αρχών σε ριζοσπαστικούς Ισλαμιστικούς κύκλους. Γίνεται αναφορά στην παραδοσιακή αρχή του που Κρύβει, αν θέλετε, τη θρησκευτική τη υπόβαθρο. Οι μουσουλμάνοι σε μη μουσουλμανικό περιβάλλον ε, μπορούν να κρύψουν τι μουσουλμανικέ του πεπιθήσει για να προωθήσουν κρυφά τον αγώνα κατά των απίστων. Πρόκειται λοιπόν για πάρα πολύ α, αφελές να θεωρήσουμε ότι οι αλλοδαποί μαχητές ή τα παιδιά τους τα οποία τα εκπαιδεύουν να γίνουν τσιγαντιστές που έχουν δολοφονήσει, έχουν βιάσει με φρικτό τρόπο. Ποιος μας εγγυάται ότι εδώ δεν μιλάμε για άτομα τα οποία θα δραστηριοποιηθούν εδώ στις επικράτειά μας και θα, επι, θα επιτεθούν στους δικούς μας. Να πω επίσης το εξής. Την εβδομάδα αυτή έχουμε το διαπίστωση την εξή, ότι οι βελγικέ αρχές δεν παρακολουθούν τους πρώην τσιχαντιστές. Τους βάζουν πέντε χρόνια φυλακή και μετά δεν παρακολουθούμε καν τι κάνουν. Θα πρέπει να κλείσουμε λοιπόν τα σύνορά μας. Ούτε τα παιδιά, ούτε οι οικογένειε τους πρέπει να γυρίσουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μα. Perdón, por el ICR, la señora Canco tiene la palabra. Thank you. I, I kept για το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Σκέφτομαι τα θύματα των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων ε, στην Ευρώπη και συνειδητοποιώ ότι μιλάμε όλο και λιγότερο για αυτά τα θύματα. Ας μην τα ξεχνάμε όμως, γιατί και αυτοί είχαν οικογένειες ε, και στις Βρυξέλλες και αλλού και ακόμα μέλη των οικογενειών και άνθρωποι που ήταν στην, στο τρομοκρατικό χτύπημα ακόμα φοβούνται να πάρουν το μετρό και ξέρετε κάθε φορά που παίρνω το μετρό και σταματάω στο Μάλμπεκ χτυπάει η καρδιά καρδιά μου και πονάει. Ε, ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λοιπόν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα θύματα. Βεβαίως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και τα παιδιά τα οποία είναι παγιδευμένα στις, ε, στη Συρία ε, και αυτά είναι ε, θύματα και, απέναντι σε αυτά τα παιδιά η συγκίνησή μου είναι μεγάλη. Βέβαια, άλλο η συγκίνηση και τα αισθήματα και άλλο η πραγματικότητα. Τα παιδιά ποτέ και με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να κληρονομήσουν τα λάθη ε, των, ε, των γονιών τους. Τα παιδιά δεν είναι ε, μόνο απειλή. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι πιο περίπλοκη από αυτήν που θέλουμε συχνά να παραδεχόμαστε. Επομένως, όλες ε, και όποιες μελλοντικές επιστροφές ε, θα πρέπει να γίνουν ε, μετά από σωστή αξιολόγηση, εντελεχή αξιολόγηση της ενδεχόμενης απειλής. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθεί και θα πρέπει να κάνουμε συζητήσεις χωρίς να υπερισχύει το συνέστημα. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία. Να μην λησμονούμε ότι η ηθαγένεια είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων υποχρεώσεων που άνδρες και γυναίκες, ε, κάποιες, ε, κάποιοι άνδρες και γυναίκες ε, παραβίασαν σκληρά. Θα πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και διακόπτεται η ομιλήτρια από την πρόεδρο. Δεν έχετε άλλο χρόνο ομιλίας. Η κυρία Νταλή έχει το λόγο. Παρακαλώ. Πολλές συζητήσεις και περιέργειες ε, έχουν γίνει εδώ, αλλά εδώ εκπλήσωμε γιατί συζητούμε εάν πρέπει ή όχι να επαναπατρίσουμε παιδιά ε, από εμπόλεμες ζώνες ε, και ότι καθόμαστε και ψηρίζουμε κατά πόσον μπορεί αυτά να αποτελούν απειλή για την Ευρώπη. Πραγματικά ε, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι α, τα καημένα αν τα αφήσουμε εκεί θα ριζοσπαστικοποιηθούν και, ή ας τα φέρουμε μόνα τους χωρίς τα παιδιά. Μα πόσα, πώς ε, ε, τολμάτε να σκέφτεστε κάτι τέτοιο. Ποιοι δημιούργησαν αυτούς τους ανθρώπους, ε, ποιοι βοήθησαν την Σύρια, πώς πιστεύετε ότι φτάσανε στην Ιράκ, στο Ιράκ και τη Σύρια, από πού ξεκινήσανε, από πού φτάσανε μέσω της Τουρκίας σε αυτά τα μέρη. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έστρεψαν κατά της κυβέρνησης του Ασάντ τους, τον Άισις και ε, ε, ε, σωστά είπε αυτός που είπε ότι αυτοί οι ξένοι μαχητές είναι ξένοι μόνο για τις χώρες τις οποίες βρίσκονται. Είναι δικά μας άτομα, είναι δικοί μας άνθρωποι. Εάν είναι τρομοκράτες, εάν φοβάστε ότι θα γίνουν τρομοκράτες, αντιμετωπίστε το. Κάντε κάτι γι' αυτό και άνθρωποι οι οποίοι ε, ε, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε «Ω Θεέ μου, έφυγαν, αποσύρθηκαν οι δυνάμεις ε, της Αμερικής από την κυρίαρχη, από τα κυρίαρχα εδάφη της Συρίας και αμάν τι έγινε». Μα τώρα το θέμα δεν είναι ανθρωπιστικό, είναι πολιτικό το θέμα και θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολιτικοί να το αντιμετωπίσουν επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στους υπόλοιπους βουλευτές που έχετε πλέον ο καθένας σας ένα λεπτό. Ένα λεπτό και θα σας κόβω το μικρόφωνο. Señor Colin Osterlet, tiene usted la palabra. Oui, madame la présidente. 700 enfants. 700 παιδιά λιγότερο των 10 χρονών ζουν σε καταβλισμούς σε Συρία σε φρικτές συνθήκες. Πρόκειται για παιδιά μαχητών. Κάθε κράτος ε, κατά περίπτωση δεν χειρίζεται τον επαναπατρισμό των υπηκόων του. Συμφωνούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πώς θα γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ποιος ε, φταίει, τα παιδιά που ε, ζουν εκεί και τι θα κάνουμε την ηλικία των 18 θα βάλουμε ως όριο για τη συγγένεια. Πώς ορίζονται τις αίματος. Πάντα ε, λέμε ότι ε, πρέπει να βλέπουμε το καλύτερο συμφέρον των παιδιών. Πρέπει να μείνουν μαζί με τις μητέρες τα παιδιά αυτά που οι περισσότερες είναι ριζοσπαστικοποιημένες. Τα κρατη τι κάνουν, τι μέτρα υπάρχουν. Όλα αυτά τα ερωτήματα δείχνουν πόσο πολύπλοκη είναι η κατάσταση πολύ διαφορετική από τη μια περίπτωση στην άλλη η κατάσταση. Πρέπει όμως να βρεθούν απαντήσεις ε, για να μην έχουμε ρολογιακές βόμβες ε, να προχωρούν ανάμεσά μας ε, αύριο. Ευχαριστώ. Παλαβρά. Thank you very much, Chair. Ο κ. Ρέσλερ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, για την θέματα ασφάλειας. Είναι προφανές ότι τα παιδιά των Ροδοπών μαχητών ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για οποιαδήποτε ασφάλματα και τις δράσεις των ε, γονέων τους. Είναι επίσης ε, σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει μία κατά περίπτωση εξέταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις και για τα άτομα τα οποία είναι σχεδόν ε, ενήλικα και για τα παιδιά. Η σύμβαση για τα παιδιά του ΟΗΕ. Θα γιορτάσουμε και την επέτειο του σύντομα. Τονίζει την ανάγκη για την προστασία των παιδιών σε τέτοιες περιπτώσει. Και να οριστεί τι είναι στο συμφέρον, προς το συμφέρον των παιδιών. Να τονίσουμε ότι υπάρχει αρμοδιότητα των κρατών μελών τα, οι πολίτε αυτοί έχουν εθνικότητα, έχουν ηθαγένεια και υπό την ε, έννοια αυτή θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κινίτση έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, ε καλεσμένους. Υπό το φως των ε, Διεθνών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού νομίζω ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί για, τον επαναπατρισμό των ε, παιδιών, των ξένων μαχητών. Πρόκειται για πολύ μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει οι ενήλικες. γνωρίζουμε επίσης ε, ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη εμπλοκή του σε τρομοκρατικές ομάδες δεν μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη. Επομένως είναι απαραίτητο να επαναπατριστούν τα παιδιά αυτά, να τους δώσουμε την απαραίτητη ψυχική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη έτσι ώστε να ξεπεράσουν το τραυματισμό τους ε, και να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία. Ε, δεν ε, βεβαίως μπορεί να είναι θέμα των μεμονωμένων κρατών μελών, αλλά δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αδιάφορη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτώ λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε ε, να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, δηλαδή να υποστηριχθούν τα κράτη ε, έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναπατρίσουν τα παιδιά τα οποία στην ουσία είναι θύματα εγκλημάτων που έχουν διαπράξει ενήλικες. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μονάχα σε επίπεδο κρατών ε, μελών μπορούν να ανακτήσουν αυτά τα χαμένα τους παιδιά. Ευχαριστώ. Fremmedkrigere er Πρόκειται για προδότες ε, που έχουν ε, προδώσει τις αρχές μας και εγώ θέλω να χαθούν. Δεν ε, θέλω να γυρίσουν. Γιατί λοιπόν άλλοι ανθρωποί μαχητές να γυρίσουν. Γιατί τι γίνεται με τα δικά μα τα δικαιώματα, με του ειρηνικού φιλήσυχου ευρωπαίου πολίτε. με το δικαίωμά μας να αισθανόμαστε ασφαλείς. Οι πολίτε αυτοί στην Ευρώπη θα πρέπει να σεβαστούν τα δικά του τα δικαιώματα πάνω από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα άλλα από μαχητών. Θα κάνω ό,τι μπορεί να από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι ποτέ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πατήσουν στο ευρωπαϊκό έδαφο. Οι Ελλαδοποί μαχητέ δεν είναι πλέον Ευρωπαίοι, είναι ο εχθρό. Δεν θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει στη χώρα μου, στην ε, Δανία και να τους ξαναμασφέρει. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ Ολλανδικά, μιας και πολλοί Ολλανδοί μιλούν Ολλανδικά σήμερα το απόγευμα. Να πω ε, ευθύ εξ αρχή το εξή. Προφανώς το θέμα αυτό προκαλεί έντονα συναισθήματα και γι' αυτό ακούμε και διάφορες απόψεις. Είναι και περίπλοκο όμως το θέμα αυτό. Περίπλοκο γιατί τα παιδιά, ένα τμήμα των παιδιών δεν αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία μας, αλλά κάποια παιδιά αποτελούν ε, κάποια στιγμή ε, από ένα σημείο και πέρα, από κάποια ηλικία και μετά 8-9 χρονών ε, ενδεχόμενο κίνδυνο για την κοινωνία μας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι έτοιμα αμφιβάλλω. Πολύ ευχαριστώ να ακούσω τι θα γίνει και στο Βέλγιο. Ίσως να έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε. Αλλά θεωρώ ότι οι κοινωνίες μας πλέον ε, δεν ε, τα αντέχουν αυτά. Το θέμα, το δεύτερο σκέλος, έχει να κάνει με τους γονείς και κατά πόσο μπορούν να συνοδεύσουν ε, τα παιδιά. Και θεωρώ ότι δεν έχουμε, δεν το ανεχόμαστε αυτό πλέον. Señora Bonviese, tiene usted la palabra. Thank you. It is precisely... Ακριβώς για λόγους ασφαλείας ε, και προς χάρη των θυμάτων είναι τόσο σημαντικό να επαναπατριστούν σήμερα αυτά τα παιδιά. Γιατί όπως φάνηκε το να μείνουν εκεί τους βοηθάμε να, ε, ε, ε να ριζοσπαστικοποιηθούν τους γονείς τους για να απαντήσουν σωστά ζητήματα ασφαλείας. Κανένα παιδί κάτω των 10 δεν ε, ποινικοποιείται. Σε κανένα κράτος μέλος, δεν διώκεται ποινικά δηλαδή. Αλλά φυσικά ε, όποιος κάνει αξιόπινες πράξεις ε, δικάζεται. Αλλά δικάζεται πού, στη χώρα του ή της. Και είναι σαφές ότι οι περισσότερες τρομακτικές απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα έρχεται από ακροδεξιούς και όχι από τον ΤΑΕΣ. και μία Βρετανίδα την οποία 15 χρονών ε, την στρατολόγησαν. Έκανε τρία παιδιά με καταναγκαστικούς γάμους σε ε, Συρία, Ιράκ και το τρίτο πέθανε ε, μετά την, τον της. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ο κύριος Σάντσεθ ήταν συντονιστής, αλλά δεν έχετε το λόγο μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Εσείς Έχετε το λόγο. Ναι, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ε, τους ομιλητές ε, και να εκφράσω την στήριξή μου στους συγγενείς των παιδιών αυτών που είναι εδώ σήμερα. Από ανθρωπιστικής πλευράς πρέπει να δράσουμε. Να δώσουμε προξενική προστασία, να επαναπατρίσουμε αυτά τα παιδιά και για λόγους ασφαλείας είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Πώς όμως να ανακόψουμε αυτές τις τάσεις ε, να αντιμετωπίζεται αυτή η απόφαση ως πολιτική. Δηλαδή υπάρχει επιλογή ε, και τελικά τα δικαστήρια ε, θα αποφασίζουν. Εκεί θα εξαρτόμαστε. Και τι μπορούμε να περιμένουμε από τις διαδικασίες στα δικαστήρια. Ακούω και κάποιους δισταγμούς και επιφυλάξεις για τον επαναπατρισμό παιδιών λόγω των γονιών τους. Η κυρία Παγάο των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να μας πει, δεν είναι και υποχρέωση των κρατών να διώκουν τους γονείς. Διακόπτεται η κυρία Στρίκ. Σενιόρ Ρος, Κύριε Ρος, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ μιλάμε για παιδιά. Και σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, μιλάμε για άτομα κάτω των 18. Μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν προσχωρήσει σε τρομοκρατικέ οργανώσει και έχουν ε, διαπράξει φρικτά εκπλήματα. Είναι ανήλικοι, αλλά, ενδια... αλλά επικίνδυνοι για την, οικογένεια, για την ε, κοινωνία μα. Γιατί να του ε, επιστρέψουμε να επανέλθουν και γιατί τους θεωρούμε θύματα, γιατί έχουμε την ψευδέστηση ότι μπορούμε να τα επιλύσουμε όλα. Το πάνελ πώς ε, τοποθετείτε με την τοποθέτηση των, ε, των ατόμων αυτών σε ε, ανάδοχες οικογένειες. Στο Άμστερνταμ είχαμε ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και τότε είχαμε πει, όταν απέτυχε το σύστημα αυτό, είχαμε πει ότι όσο εδώ και μη παρέκει, αλλά πάντα επιτρέπουμε και παραπάνω. Αλλά βασικό μας καθήκον είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Γι' αυτό έχουμε εκλεγεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μπάλας. Πώ Πώς να σκεφτεί καν κανείς ότι θα αποχωρήσει τα παιδιά από τους γονείς τους. Θυμάμαι τι έγινε ε, στην Ιρλανδία όταν έπαιρνε από τις ανήπαντρες μητέρες η Καθολική Εκκλησία τα παιδιά τους. Πότε θα αναλάβει την ευθύνη της η Ευρώπη για τις ασφερκαλαιότητες που ήδη έχει προκαλέσει στη Συρία. Έχουμε ξεχάσει ότι εξοπλίσαμε τους τζιχαντιστές και ότι πυροδοτήσατε την ε, ε, ανατροπή όλων αυτών των καθεστώτων και αυτό που ε, επακολούθησε. Βοηθήσατε να πέφτουν βόμβες στα παιδιά ε, και στα, στις στέγες των σπιτιών τους και τώρα σας νοιάζει τι γίνεται σήμερα ε, στο Ιράκ, στην Ιεμένη ε, τι σας ε, νοιάζει, τι γίνεται εκεί πέρα, σε τι πλανήτη ζούμε πλέον. Ευχαριστώ. Κυρία Φόξ τώρα. This is an Είναι σημαντικό το θέμα και είναι περίπλοκο ηθικά και γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να το επιλύσουν να τα επιλύσουμε σε, με κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις. Αν ήταν θέμα Ευρωπαϊκή Επικυριαρχία, Εθνική Επικυριαρχία, είναι το κατεξοχήν θέμα Εθνική Επικυριαρχία. Γιατί αυτό σχετίζεται με του Ευρωπαίου πολίτε και τα δικαιώματά του και πώ αντιμετωπίζουμε του ε, συμπολίτε που πρόδωσαν τι αξίε του και γύρισαν την πλάτη του Στον ανθρωπισμό και την ε, δυτικό πολιτισμό. Η Βρετανική κυβέρνηση αρνήθηκε επαναπατρισμό σε περίπτωση συγκεκριμένη. Πιστεύω ότι ήταν λάθο και ήταν δειλία αυτή, γιατί δεν ανέλαβαν τι ευθύνε του. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνε μας. Αλλά αυτό είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το αποφασίσουν ε, οι Βρετανοί πολίτες, όχι να επιβληθεί από πάνω από τη γραφειοκρατική Ευρώπη. Χρησιμοποιούνται λοιπόν τεχνικές για να εκβιάσουν τα κράτη-μέλη, για να επιστραφούν οι μητέρες των πετρελαίων αυτών. Ευχαριστώ πολύ και διακόπτει ο Πρόεδρος. Wesley Lima. Καταρχάς να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο για να εξηγήσουν αυτό που συμβαίνει και να εκφράσουν απόψεις. του δύο ερωτήσει έχω. Η πρώτη είναι τι έγινε από τι χώρε που επαναπάτρεσαν τα παιδιά. Τι υποστήριξη είχαν αυτά τα παιδιά. Δεύτερον, να μην έχουμε μόνο παραδείγματα, αλλά για το πάνελ συγκεκριμένα, σε όλα τα μέλη στρέφομαι τώρα, ε, κάποιες ε, διαδικασίες, δηλαδή να δούμε την, ίδια, την όλη διαδρομή, κάποια στοιχεία ε, που να συνιστούν αυτή την επιτυχία. Να δείξετε δηλαδή ότι είναι μια επιτυχημένη προσέγγιση, γιατί μόνο έτσι τέλος πάνω, με τον αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να πείσουμε όσους δεν πείθονται εύκολα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος όλες και όλους και λυπούμε πολύ που σε κάποιους χρειάστηκε να κόψω το μικρόφωνο. Θα σας είχα δώσει και δύο και τρία και τέσσερα λεπτά αν μπορούσα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα. Έχετε τώρα παρακαλώ εσείς του πάνελ 6 λεπτά ο καθένας, αλλά θα είμαι και με εσάς εξισουαστήρι, όσο και με τους βουλευτές. Να ξεκινήσουμε με τη σειρά ε, την αντίθετη αυτή τη φορά, άρα θα δώσω καταρχάς το λόγο στην κυρία Χέν. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η συζήτηση πραγματικά αυτή είναι πολύ έντονη και το θέμα αυτό έχει προκαλέσει έντονα τραύματα σε όλους τους Ευρωπαίους. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα η συζήτηση να επανέλθει στα παιδιά. Το γεγονός ότι η προσελκυσμός των παιδιών από τέτοιε ενόπλε ομάδε, όποιε να είναι αυτές οι ενόπλε ομάδε, αποτελεί μεγάλη παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών υπό το διεθνέ δίκαιο. Και έχουμε προγράμματα και μηχανισμούς για να επανεντάξουμε τα παιδιά αυτά. Είτε είναι παιδιά στη Συρία, είτε είναι παιδιά στη Βυτική Αφρική, τα παιδιά αυτά είναι θύματα και υπάρχουν προγράμματα επανένταξη για τα, για τα παιδιά αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναμπούν στην κοινωνία και αυτό ξεκινά με την οικογένειά τους. Δεν θα θέλαμε να μπουν σε ιδρύματα τα παιδιά αυτά. Η φροντίδα στους κόλπους της οικογένειας είναι πάντα η καλύτερη δυνατή λύση για την υποστήριξη έχουμε κυβερνήσεις που παίρνουν ε, τα παιδιά αυτά πίσω, τα επιστρέφουν, τα επαναπατρίζουν. Το Κόσοβο, για παράδειγμα, 70 παιδιά πήρε. Και α είμαστε ρεαλιστέ, τα παιδιά αυτά θα αποτελέσουν μια ομάδα η οποία θα απαιτήσει πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να μπορέσουν να συνέλθουν κατά κάποιο τρόπο από αυτά που συνέβησαν. Άλλα κράτη-μέλη επίση εργάζονται από αυτόν. 380 άτομα επίστρεψαν στην ε, Βρετανία. βάσει της ε, έκθεσης για τη στρατηγική της Μεγάλης Βρετανίας ε, σε ό,τι αφορά το κατά πόσο αποτελούν ε, απειλή τα άτομα αυτά. Η κυβέρνηση ξέρει που βρίσκονται, τα παρακολουθεί, είναι σε επαφή μαζί τους. Έχουμε και μια ανθρωπιστική οργάνωση. Δεν εξετάζουμε θέματα που αφορούν καθαρά την ασφάλεια και τις απειλές, αλλά σημειώνουμε ρυθμιστικές υπηρεσίες δύο κρατών μελών της Ολλανδίας και της Σουηδίας έχουν ε, εκφέρει την άποψη ότι οι οικογένειες που επαναπατρίζονται, μιλώ για οικογένειες, όχι για παιδιά, είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας. Οι μητέρες και τα παιδιά νομίζω ότι είναι σε άλλη κατηγορία. Αυτό είναι σαφές. Είναι πολλοί που έχουν μετανιώσει και το μόνο που θέλουν είναι να πάνε σπίτι τους. Κάποιοι άλλοι διατείνονται ότι είναι φυλακισμένοι εκεί και θα προτιμούσαν να είναι σε φυλακή στην πατρίδα τους τουλάχιστον προκειμένου τα παιδιά τους να είναι με την οικογένειά τους. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θα πω. Θέλω να τονίσω πόσο κατεπήγουν είναι ο χαρακτήρας των ανθρώπων αυτών. Μιλάμε για εξέταση κατά περίπτωση οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και αυτό ενδεχομένως ε, να μην το συζητάμε πλέον από το νέο έτος. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα πάρουμε τα παιδιά αυτά και τους στενούς συγγενείς τους και να τους βγάλουμε από την κατάσταση αυτή που βρίσκονται σήμερα. Δεν μπορώ να το πω με άλλα λόγια. Πρέπει να συμφωνήσω με τον συνάδελφο στο πάνελ. Μιλάμε με ωραία λόγια, αλλά χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών και έχουμε τη δυνατότητα για να βγάλουμε τα παιδιά αυτά από εκεί. Τώρα θα πρέπει να ενεργήσουμε η έλλειψη δράσης, η μη ανάληψη δράσης θα είναι θαντική καταδίκη για τα παιδιά αυτά. Το υπογραμμίζω αυτό. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να κοιτάξουμε τι γίνεται κατά περίπτωση στη Συρία. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα παιδιά αυτά. Τώρα χρειαζόμαστε όμως μια συνολική λύση και μετά θα κοιτάξουμε κατά περίπτωση τι γίνεται. Τα κρατημέλη λοιπόν θα πρέπει να προτείνουν επαναπατρισμό στα παιδιά αυτά, σε όλα τα παιδιά αυτά και στι οικογένειε του, στι μητέρε του στο σύντομα των δυνατών. Ευχαριστώ, όπως είπα, πάμε με την αντίθετη σειρά αυτή τη φορά, οπότε τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βαν Τίχελτ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να δώσω κάποιες απαντήσεις. Ακούσαμε τις ερωτήσεις και τις διάφορες προοπτικές, συναισθηματική, ανθρωπιστική, γεωπολιτική, δικαστική, οπτική διεθνούς δικαίου και το καθεξής. Η δική μου είναι βέβαια πιο πολύ η πτυχή της ασφάλειας. Αυτή είναι η οπτική ε, η δική μου πιο πολύ και πάνω σε αυτό να απαντήσω τις ερωτήσεις. Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Κοιτάξτε, όλοι οι ενήλικοι, για τους ενήλικους μιλάω τώρα, φυσικά και πρέπει να δικαστούν, να ε, αυτό που λέμε προσέγγιση ποινική δικαιοσύνη. Είναι ξεκάθαρο στη χώρα μου αυτό. Το ίδιο ισχύει για τι γυναίκε. Πολλέ έχουν καταδικαστεί και μάλιστα ειρήνη. Θα μπορούσαμε να το, έχουμε, να το συζητήσουμε και το συζητούμε και γι' αυτό υπάρχουν τα κοινοβούλια. Μπορούμε να μιλάμε για το κατά πόσο μια ποινή κράτηση αρκεί πέντε χρόνια. Δεν ξέρω, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση. Να την κάνουμε, δεν λέω, αλλά είναι σημαντική η προσέγγιση ποινική δικαιοσύνη. Στην πράξη, τι θα πει. Όταν εγώ σπούδαζα νομική ε, σημαίνει adjudicare, λαμβάνοντας όλες τις προοπτικές. Δικάζονται στη χώρα καταγωγής ή στη χώρα που διέπραξαν ε, την αξιόπινη πράξη. Αν δικάζονται στη χώρα που ε, διέπραξαν την αξιόπινη πράξη, το ξέρουμε, αν και δεν μας αρέσει, ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν τα πρακτικά και τα νομικά εμπόδια. Όσο δε περισσότερο το συζητούμε, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν να δικαστούν εκεί πέρα. Από την πλευρά της ασφάλειας τώρα. Πάντα. πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τις γυναίκες, ε, ε, τα στρατόπεδα για τους άντρες φυλακές. Ε, τέλος πάντων υπάρχει ο κίνδυνος να ξαναστρατολογηθούν από τζιχαντιστές, είτε είναι σε στρόπεδο είτε είναι σε φυλακή. Πάντα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αναπτύξουν αισθήματα μίσους σε βάρος της δύση. Δεν, έχουν την δεν έχουν την ευθύνη και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο αυξάνουν τα αισθήματα μίσους. Και ακόμη και όταν κανονικά θα έπρεπε να μπορούμε, πρέπει να τους δικάσουμε στο Ιράκ, με βάση τις αρχές μιας δίκης δίκης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ταυτόχρονα τον κίνδυνο να απελευθερωθούν ξανά. Αυτή είναι η μακροπρόθεσμη προοπτική. Εγώ έχω το καθήκον να προειδοποιώ τις αρχές με βάση τη δική μου οπτική. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τι που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όταν θα φεθούν ελεύθεροι. Ξέρετε τι έγινε στο Ghraib και στην Baghdadi και άλλοι ε, συναντήθηκαν και ε, ανέπτυξαν σε αυτές τις φυλακές ακριβώς τα αισθήματα μίσου, φυλακές του Ιράκ. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όπως και τον αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις μας σε οικογένειες ε, εδώ, ε, στις κοινότητες εδώ, στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να δοθεί η αίσθηση εγκατάλειψης, ούτε της δημιουργίας κατηγο... δεύτερη κατηγορία πολιτών. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Έχω 6 λεπτά, δεν μου είπατε. Α, δύο εννοούμε. μου Πάει ανάποδα το χρονόμετρο, μάλιστα. Από βελγικής πλευράς έχουμε 130 ενηλίκους που επιστράφηκαν Τα καμία τρια παιδιά, τα βάζουμε στη φυλακή, τα, απελευθερω... τα βγάζουμε έξω και μετά τα παρακολουθούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγγύηση δεν υπάρχει όμως, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν υπάρχει ο μηδενικός κίνδυνος. Ό,τι και αν κάνουμε, είτε εδώ είτε εκεί, υπάρχει κίνδυνος. Το ο μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει, ας το χωνέψουμε, ακόμη και αν δεν μας αρέσει. Και με τα δικά μου τα παιδιά, που δεν έχουν πάει ποτέ εκεί. Έχω εγώ εγγύηση ότι θα τους δώσω τη σωστή ανατροφή, παρότι, να σας διαβεβαιώσω, είμαι πολύ καλός πατέρας, έτσι Λοιπόν, δεν υπάρχει μηδενικό κίνδυνο όμω επαναλαμβάνω. Υπάρχει παρέμβαση ενός ε, μελτή ανηλίκων ε, που αναλαμβάνει τα παιδιά. Υπάρχουν υπηρεσίες πρόνοιας και άλλες δομές στη χώρα μου. Έχουμε πραγματικά πραγματική δέσμευση αυτών των δομών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξαναπάνε σχολείο τα παιδιά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Είναι η υποχρέωσή μας. Παναλαμβάνω όμως, εγγύηση δεν υπάρχει ε, για την επιτυχία. Για το χρονοδιάγραμμα που λέγει ο κύριος ε, Πέτερς, τέλος πάντων το, το παράθυρο, το χρονικό σας είπα, όσο περισσότερο περιμένουμε, ε, τόσο περισσότερο κινδυνεύει να δημιουργηθεί μια νέα γενιά τζιχαντιστών. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση από ανθρωπιστική πλευρά και με τι τελευταίε εξελίξει η κατάσταση έγινε πολύ χειρότερη και από πλευρά ασφαλεία. Είναι και πιο δύσκολο τώρα δηλαδή οι δυτικέ δυνάμει να επαναπατρίσουν τα παιδιά του. Κάποιοι σύμμαχοι και φίλοι αποσύρονται από εκεί. Άρα όλα αυτά δεν διευκόλυναν την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθειά σας. Ο κύριος Μαρτίν δεν ήταν εδώ όταν ε, παρενέβη ε, συντονιστής από την ομάδα σας κάποιος άλλος, αλλά έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας αν θέλετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πραγματικά το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ε, καυτό και πολύ περίπλοκο. Και δυστυχώς ε, είναι λυπηρή η κατάσταση αυτή για τα μικρά παιδιά. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα αυτό όχι μόνο από ηθικής πλευράς, γιατί και η πολίτες των κρατών μελών ε, έχουν δικαίωμα να, μην, να έχουν ένα ασφαλής. Πολλοί λοιπόν είναι, ε, έχουν υποστεί τραύματα, αλλά έχουν διαποτιστεί και από την προπαγάνδα του ίσης και επιστρέφουν λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις ε, στις χώρες μας εδώ και στη Γερμανία. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ασφαλείας και να ελέγχεται από τις σχετικές υπηρεσίες τι γίνεται και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σωστοί όροι να αφαιρείται το δικαίωμα και δαιμονία του. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν στην Ευρώπη περαιτέρω τζιχαντιστές, μαχητές. Παρακαλώ ησυχία στην αίθουσα, λέει η πρόεδρος. Η κυρία Χένα έχει το λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτήν τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις ε, Νομίζω ότι η συζήτηση κατέδειξε και το περίπλοκο του ε, θέματος, όπως ο Πολ Φαντίχελτ ε, ήδη είπε. Ε, εξεφράστηκαν απόψεις επί πολλών ζητημάτων. Παρ' όλα αυτά ε, κατεδείχθη σαφώς ότι ούτε τα ερωτήματα είναι εύκολα, ούτε και οι απαντήσεις τους. Κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά και κάποιες ε, προειδοποιήσεις όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον, κατά πόσον μπορεί να συμβάλλει στην επιστροφή ε, παιδιών. Ε, αυτά είναι εθνικά ζητήματα και αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η κατάσταση. Όπως όμως υπόθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διευθετήσει κάποια ζητήματα τα οποία ηγέρθησαν εδώ στη διάρκεια της συζητήσεως. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανταλλαγή απόψεων λοιπόν, και πληροφοριών σχετικά με το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Ένα σημαντικό ζήτημα και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι εδώ το ε, αναφέρθηκαν ε, στην ασφάλεια των συνόρων, δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι όταν κάποιος μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αν πρόκειται για να ανοιχνεύεται και να ταυτοποιείται αν και εφόσον είναι είτε ο ίδιος ξένος μαχητής είτε μέλος της οικογένειας κτλ. Έχουμε πληροφορίες λοιπόν και θέλουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες ε, ε, και τις πληροφορίες που παίρνουμε από τις Πολιτείες, από την Ίντερπολ που αφορούν Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο σημαντικός ρόλος που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να διασφαλίσει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την ανταλλαγή πληροφορών είναι η Europol. Ε, είχαν την πρώτη task force για την ε, ταυτοποίηση τρομοκρατών και προσπαθούν να φέρουν ε, οι εμπειρογνώμονες διαφόρων χωρών γύρω από το τραπέζι έτσι ώστε να συγκρίνουν στοιχεία και πληροφορίες για να έχουν κάποιες, κάποια νέα στοιχεία. Όσον αφορά τις καλές πρακτικές, σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, την αποκατάσταση ε, και γενικότερα συνοδεύει τις χώρες ε, ε, σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης, ας πούμε, μέσω του δικτύου που έχουν δημιουργήσει οι εμπλεκόμενοι με το θέμα. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η Πρόεδρος, κυρία Παρόν, ε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για το βάθος ε, αυτής της ε, συζήτησής μας σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι αυτή η συζήτηση αφορά θέματα πολιτικά, θέματα ασφαλείας και άλλα και κοινωνικά. Δεν είναι αφελές να πει κανείς ε, ότι ο επαναπατρισμός ε, έχει και περιλαμβάνει και στοιχεία ασφάλειας. Ε, το θέμα του, των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και αντικατοπτρίζεται και στην συνολική στρατηγική κατά της τρομοκρατίας. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία απέναντι στα θύματα. Όσοι έχουν ε, εμπλακεί σε ε, τρομοκρατία θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν από δίκη. Και εάν εμείς αφήσουμε αυτούς που δραπετεύουν από τα στρατόπεδα, έτσι όπως έχει κατάσταση σήμερα ε, στην ε, βορειοανατολική Συρία, όπου είναι ιδιαίτερα ρευστή η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια, εάν τους επιτρέψουμε να εξαφανιστούν και να τους χάσουμε, αυτό στην ουσία ε, δείχνει μη σεβασμό για τα θύματα. Επίσης ε, θα πρέπει και τα θύματα να έχουν τη δυνατότητα να ακουστούν. Ας πούμε στις δίκες ε, που ξεκίνησαν στο Ιράκ ε, για, τον, για την τρομοκρατία, εκεί δεν υπάρχει θέση για τα θύματα. Είναι συνοπτικές οι διαδικασίες, είναι γρήγορες, πολύ γρήγορες οι δίκες και οι ενώσεις των θυμάτων δεν είχαν τη δυνατότητα ε, να ακουστούν. Επομένως, η λογοδοσία ε, απέναντι στα θύματα είναι ε, επίσης κάτι σημαντικό. Είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε ενώπιν της δικαιοσύνης όσους έχουν διαπράξει αδικήματα αλλά η ποινική ευθύνη είναι ατομική και επομένως δεν είναι δυνατόν να βάζουμε όλους στο ίδιο καλάθι, όπως είπε προηγουμένως ένα συνάδελφος. Θα πρέπει να γίνει ένα screening σε ε, επίπεδο ε, ατομικό να δούμε κατά πόσον ένα άτομο είναι υπεύθυνο και αν είναι υπεύθυνο για εγκληματικές πράξεις και για αδικήματα τότε να περάσει από ε, δίκη. Δεν υπάρχει λόγος αντικατάστασης ε, για ε, χώρες οι οποίες έχουν δικαϊκό σύστημα σωστό κτλ. Αυτή, αυτά τα συστήματα οπωσδήποτε όσους έχουν διαπράξει αδικήματα θα τους φέρνουν αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ε, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά. Η UNICEF μεταξύ ε, εντός του συστήματος του ΟΗΕ έχει μακρά πείρα εργασίας με αυτά τα παιδιά, με παιδιά στρατιώτες ε, παιδιά που έχουν εμπλακεί σε ε, επιθέσεις και πολέμους. Το πώς δηλαδή ε, ξαναπάμε τα παιδιά αυτά στο σχολείο, πώς ε, τα ξαναεντάσσουμε στην κοινωνία. Υπάρχουν κυβερνητικές οργανώσεις ε, που δουλεύουν εντός των κρατών μελών, που μπορούν να ενδυναμώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν κατά την έννοια αυτή. Υπάρχει η UNICEF λοιπόν και βοηθούνται όλοι αυτοί από τη UNICEF. supports uh, all requests coming from member Thank you very much. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εισηγητές για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει. Ε, ε καταλαβαίνω ότι αυτά που υπόθηκαν εδώ ε, είναι σημαντικά ε, και τα, και τα δικαιώματα είναι αναπαλωτρίωτα αλλά και οι υποχρεώσεις και δεν θέλουμε ατιμορρησία σε οποιαδήποτε ε, περίπτωση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τιμωρηθούν αυτοί που φέρουν ευθύνες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες ε, και να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι στις 20 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα μία υψηλού επίπεδου διάσκεψη ακριβώς για τα δικαιώματα των παιδιών. Ε, αυτή η διάσκεψη σηματοδοτεί το, ε, την 60η επέτειο της δήλωσης για τα δικαιώματα των παιδιών των Ηνωμένων Εθνών καθώς επίσης και την 30η επέτειο της Σύμβασης για τα δικαιώματα δικαιώματα των παιδιών. Ε, επιθυμίζουμε με την διοργάνωση αυτή τη σημαντική διάσκεψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί ε, να είναι δεσμευμένο στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Ε, εκεί θα συζητήσουμε λοιπόν εν μέρει αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Let's start, colleagues. Преминаваме към точка 22, доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета за напред. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να περάσουμε στο σημείο 22. Έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο τη Βουλγαρία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασία και Ελέγχου. Και το σημείο 23 σε ό,τι αφορά ε, την περίπτωση της Ρουμανίας, την πρόοδο της Ρουμανίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 22 Οκτωβρίου του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο εκθέσεις για την πρόοδο της Βουλγαρίας και την πρόοδο της ε, Ρουμανίας ε, υπό τα πλαίσια του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου. Αυτός ο μηχανισμός δημιουργήθηκε με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007 και ήταν ε, προσωρινός μηχανισμός προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια των δύο χωρών να μεταρρυθμίσουν ε, το δικαστικό τους ε, τομέα και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματο σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η πρόοδο που έγινε από τη Βουλγαρία στάση του μηχανισμού είναι επαρκής για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι έχουν τηρηθεί μεύσεις της Βουλγαρίας. Ε, φυσικά, η Βουλγαρία θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την συνεχιζόμενη εφαρμογή της μεταρρύθμισης ε, και όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη στους μελλοντικούς διαλόγους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού του κράτους δικαίου. Σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία, Η έκθεση σημειώνει ότι η εξέλιξη της κατάστασης της πρώτης μήνες του 2019 ήταν ε, πηγή μεγάλης ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ρουμανία δεν ε, ε, δεσμεύτηκε σε διαφορά τη τις επιπρόσθετες συστάσεις που έγινε τον Νοέμβριο του 2018 που ήταν όμως κοινέ από, την, από όλα τα θεσμικά όργανα. Θα δώσω το λόγο στο William Σλίθ, ο οποίο είναι ε, διευθυντή για του πολίτε, τη μετανάστευση και την Ένωση Ασφάλεια από τη Γενική Γραμματεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μα παρουσιάσει τα πορίσματα των δύο αυτών εκθέσεων. Κύριε Σλίθ έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις δύο εκθέσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού CVM. Ενδεχομένως να σας βοηθήσω, να σας το πλαίσιο. Ο μηχανισμός αυτός ήταν ένας μηχανισμός ε, ο οποίος ήταν ο μακρυπρόθεσμος όταν ε, προσχώρησαν τα διευτα κρατη κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέλαβαν κάποιες δεσμεύσεις για το πώς θα τηρηθούν ε, οι δεσμεύσει αυτέ περιληφθήκε σε κάποιε αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιανουάριο του 2017, λοιπόν, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια δεκαετή έκθεση για το πώ πάνε τα πράγματα, για να μα δώσει μια συνοπτική ε, θεώρηση τη περίοδου αυτή. Ω αποτέλεσμα, εστιαστήκαμε καταρχά σε ένα περιορισμένο αριθμό βασικών συστάσεων για να δούμε τα βήματα που χρειάζονται σε βασικούς τομείς και κάποιες προκλήσεις για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και κατά δεύτερον, μία, ένα κάποιον έλεγχο, γιατί φυσικά οι εξελίξεις και η πρόοδος δεν σημαίνει ότι έχουν τραπεί τάσεις που είχαν παρατηρηθεί. Έχουμε επικεντρωθεί λοιπόν σε δύο τέτοια ερωτήματα. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την προθυμία της να κάνει άλλη μία έκθεση πριν το τέλος ε, της θητείας. Όπως ε, είπε και ο Πρόεδρος, τα δύο αυτά θέματα θα κοιτάξω από κοινού. Θα ξεκινήσουμε όμως με τη Βουλγαρία. Από τον Ιανουάριο του 2017 οι εκθέσεις έχουν εντοπίσει σαφή πρόοδο Πέρσι έκλεισαν τρία ορόσημα, για παράδειγμα. Βασικά βήματα για την νομική διαδικασία ήταν ε, μια νέα υπηρεσία κατά της διαφθοράς, ε, νέες αρμοδιότητες για ιστορικούς ελέγχους και αλλαγές ε, στις ποινικέ διαδικασίες κατά τη διαφθοράς, συνεργασία η οποία συνεχίστηκε έκτοτε και η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Βουλγαρία συνεχίζει να εργάζεται για την εφαρμογή των συστάσεων του τελευταίου έτος, σημειώνοντας περαιτέρω πρόοδο και σε ό,τι αφορά τη σύσταση για την ολοκληρώση των τριών σήμων benchmarks που ολοκληρώθηκαν πέρσι για τη διαφθορά. Και συμπερασματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπέρανε ότι με τα βήματα που έγιναν για τις μελλοντικές πρόοδους. Η πρόοδος που σημείωσε η Βουλγαρία υπό το μηχανισμό CVM ήταν επαρκής. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλγαρία θα μπορούσε να περάσει στο νέο καθεστώς ένα μηχανισμό κράτους δικαίου και τις πολιτικές καταθυντήριες για το επόμενο διάστημα, όπως ε, ορίστηκε και στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι τον Ιούλιο. Αυτό θα σημαίνει διάλογο με όλα τα κρατημέλη, με έναν ετήσιο κύκλο υποβολή αναφορών για να κοιτάξουμε θέματα που άπτονται του κράτου δικαίου. Να υπενθυμίσω ότι οι συστάσει του CVM δεν τα καλύπτουν όλα, μόνο τα θέματα που είχαν εντοπιστεί στην αρχή της διαδικασίας. εντοπίζεται το ευρύτερο πλαίσιο. Το νέο Συμβούλιο Συνεργασίας, λοιπόν, το οποίο ιδρύθηκε στην Βουλγαρία, όχι μόνο θα είναι ο βασικός εθνικός φορέας για τέτοια θέματα, αλλά και σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά και τα άλλα θεσμικά όργανα εξακολουθούν να έχουν ρόλο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το δικαστικό σώμα, το οποίο προασπίζει τους δικαστές και όλα αυτά θα αποτελέσουν και στο μέλλον εξίσου σημαντικά όργανα, όπως και σήμερα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την έκθεση, αλλά θα ήθελα να ε, πω ότι υπάρχουν τέσσερις συγκεκριμένε δεσμεύσεις από πλευρά των βουλγαρικών αρχών τονίζονται αυτά στο τέλο τη έκθεση. Καταρχάς, στο ευαίσθητο θέμα της λογοδοσίας του Γενικού Εισαγγελέα. Η ε, Βουλγαρία έχει γράψει στην Επιτροπή της Βενετίας και έχει ακολουθήσει τις συστάσεις αυτές ε, σε, ό,τι αφορά φυσικά και τους περιορισμούς που, του συντάγματος της Βουλγαρίας. Κατά δεύτερον, η Βουλή έχει εξετάσει το πώς θα απαλληλθούν οι ανησυχίε για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Κατά τρίτον, η βουλγαρική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να συνεχίσει με το, τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για το πλαίσιο κατά της διαφθοράς και για να είναι αποτελεσματικές οι ποινικές μελέτες. Η Επιτροπή λοιπόν διαπιστώνει ότι έχει πληρώσει τους όρους που χρειάζεται η Βουλγαρία. Αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να τοποθετηθούν. Θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη προτού επίσημα τερματιστεί ο μηχανισμός CVM για τη Βουλγαρία. Τώρα να κοιτάξουμε τη Ρουμανία την τελευταία έκθεση τον Νοέμβριο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπέρανε ότι οι εξελίξει ε, στην Ρουμανία είχαν κάνει πίσω σε ό,τι αφορά την πρόοδο. Για παράδειγμα, ε, τα νομοσχέδια για τη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά και την τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτό δεν αποτέλεσε μονομένη άποψη. Ήταν ε, σε αρμονία και με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και με τα απορίσματα της ε, Επιτροπής της Βενετίας. Ήταν ομόφωνη λοιπόν η άποψη όλων των ε, οργάνων αυτών. Έκανε λοιπόν οκτώ επιπλέον συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρα από αυτές που είχαμε κάνει το 2017. Δυστυχώς δεν ακολουθήθηκαν αυτές οι συστάσεις και του μήνες μετά την ε, έκθεση υπήρχαν περαιτέρω περιστατικά που επιδίνωσαν την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέφυγε στις ρουμανικέ αρχέ σε διάφορες περιστάσεις. Έγραψε μια επιστολή, για παράδειγμα, για, ανησυχία, για ανησυχίες για το κράτο δικαίου, το Μάιο. Ωστότε ήταν αρνητικές οι δράσεις ε, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να ε, υπάρξει εναστατικός χαρακτήρας, δεν έχουν επιληθεί ακόμα τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια για το δικαστικό, για το ποινικό δίκαιο και για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος. Σε κάποιες περιστάσει, οι επιπρόσθετες συστάσει του Νοεμβρίου του 2018 δεν έχουν ουσιαστικά εφαρμοστεί ακόμα και οι ανησυχίε εξακολουθούν να υφίστανται. Η εμπειρία μας από τον Νοέμβριο του 2018 έχει επιβεβαιώσει τις ανησυχίες μας. Έχουμε λοιπόν επιπλέον λόγους ε, που να δικαιολογούν ε, τους φόβους μας. Κίνδυνος λοιπόν πολιτικής ανάμειξης. Δεν υπάρχει ένδειξη στην παρούσα φάση ότι θα υπάρξει διαβούλευση με την Επιτροπή της Βενετίας. Και οι δράσεις ελέγχου μας έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω ανησυχίε. Πίεση, για παράδειγμα, υπάρχει όλο και περισσότερη για τον εισαγγελέα, για το δικαστικό σώμα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά η γενικότερη πολιτική δεν έχει αλλάξει. Η πρώτος τώρα σε σχέση με τις συστάσεις του 2017 ήταν και αυτή αργή. Πολλά από αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με τη σαφήνεια, τη διαβούλευση και τη συνεργασία. Και πολλά από αυτά πάνε πίσω. Σε κάποιους τομείς, όπως ε, συστήματα για τις δημόσιες προμήθειες ή για, την, ε, για τα περιουσιακά στοιχεία. Εδώ έχει σημειωθεί πρόοδος. Αλλά και πάλι άλλες εξελίξεις δεν ε, θεωρούμε ότι έχουν ε, προωθήσει τις συστάσεις. Άρα θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι συστάσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ρουμανικές αρχές προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σλίτ, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ενημερώσω πως σήμερα και αύριο η Επιτροπή Βενετίας συνεδριάζει στη Σόφια για να έρθει σε επαφές με τις αρχές εκεί και να βαληθεύσει όλα αυτά τα που μας ανέφερε η Κομισιόν. Τώρα, θα ήθελα να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων, δεν υπάρχει πολύ χρόνος, οπότε δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε τα δύο λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές και πρώτην κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ πολύ. Το ΕΛΚ στηρίζει τα συμπεράσματα της Κομισιόν και συμφωνεί σε ό,τι αφορά την πρόοδο της Βουλγαρίας του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου. Άρα πληρούνται οι δεσμεύσεις της για προσχώρηση στη, ε, ε, στο μηχανισμό, στο χώρο του Σέγγεν. Και πρέπει να λήξει η συμμετοχή στο μηχανισμό. Το 2007 ε, εντάχθηκε σε αυτό το μηχανισμό για να επιταχυνθούν οι προσπάθειες της χώρας ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος και βελτίωση της καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς. Η εκτίμηση τη πρόοδου τη Βουλγαρία από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά αυτό το μηχανισμό περιλαμβάνει κάποια κριτήρια. Το Νοέμβριο του 2018 είχαν ε, ήταν θετική η ανταπόκριση χώρα σε αυτά τα κριτήρια, νομοθετικέ διαρθρωτικές αλλαγέ ε, ευθυγραμμίζονται με το μηχανισμό. Αποφασίστηκε τότε βέβαια να ε, ξαναγίνει ε, έκθεση. Με την τελευταία αυτή έκθεση πρόοδου βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά όλα τα κριτήρια πλέον είναι ικανοποιητική η απόδοση της Βουλγαρίας. Έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες η χώρα στους τομείς αυτούς. Έχει τοποθετηθεί ε, και η Κομισιόν και πιστεύω ότι το κλείσιμο αυτού του μηχανισμού είναι ένα θετικό μήνυμα και προς το λαό της χώρας. Μία υποσημείωση όμως, αν όπως αναφέρθηκε θέλουμε να έχουμε ένα εργαλείο παρακολούθησης του κράτου δικαίου που θα βλέπετε κειμενικά την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη. κάτι το οποίο ζητάμε άλλωστε εμεί στο Κοινοβούλιο εδώ και καιρό. Ίσως τότε όλος ο μηχανισμός συνεργασία και έλεγχου θα ήταν περιττός, εφόσον θα υπήρχε αυτό το συνεκτικό εργαλείο παρακολούθησης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζήπελ, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το μηχανισμό συνεργασίας και έλεγχο για τις δύο χώρες. Αλλά θα υπογραμμίσω όπως και η Ρομπέρτα Μέτσολα ότι και εμείς, το, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, ζητούμε να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός παρακολούθησης του κράτους δικαίου Δηλαδή, έχει νόημα να έχουμε μηχανισμό που θα εφαρμόζεται σε μεμονωμένα κράτη, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να υπάρχουν ήδη κανόνες για όλα τα κράτη. Εξού λοιπόν και ζητώ ένα νέο μηχανισμό για το κράτος δικαίου που θα οδηγήσει σε ακύρωση, δεν θα είναι πλέον δηλαδή, θα είναι πια περιττός αυτός ο μηχανισμός CVM, μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου. Θέλουμε επίσης ε, να χαιρετήσουμε το κλείσιμο του μηχανισμού για την ε, Βουλγαρία και να αναφέρουμε κάτι ακόμη. Το χώρο του Σέγγεν πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως ε, το κεκτημένο Σέγγεν που δεν έχει άμεση σχέση ακριβώς με το μηχανισμό συνεργασία και αν έχουμε την έννοια ότι θα πρέπει να αρθούν πλήρως οι απαιτήσει και υποχρεώσει για την ε, εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν από την Βουλγαρία και οι δύο χώρες, Βουλγαρία και Ρουμανία. Άλλωστε μπορούν να πληρούν τις ε, προποθέσει για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν. Τα λέμε αυτά στι εκθέσει μα. Έκθεση 2 πρωτοβουλία του Δεκεμβρίου 18 τελευταία. Που ζητούμε και θυμίζουμε την πλήρη εφαρμογή του Σέγγεν, λέγοντα ότι δεν εξαρτάται από το μηχανισμό. Άρα, ζητούμε ίσως όχι από την Κομισιόν, από τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, αυτό που πρέπει ώστε Βουλγαρία και η Ρουμανία να γίνουν πλήρη μέλη του χώρου Σέγγεν. Και σε ό,τι αφορά το CVM πρέπει να σταματήσει να ισχύει, να καταργηθεί και να βρεθεί πλέον ένας μηχανισμός ε, που θα ελέγχει με πολύ φιλικό τρόπο όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στράικ. Sorry, I was waiting for renew. ναι, νόμιζα ότι θα δίνετε πρώτο το λόγο στον εκπρόσωπο του Renew. Thank you. Um, on behalf of Renew... Εξ ονόματος ε, του, ε, της ομάδας ε, Renew, uh, θα αποφάσισα να μιλήσω στα ε, αγγλικά, ενώ αρχικά είχα πει να τα πω ρουμάνικα ως ε, Ρουμάνος, αλλά είμαι συντονιστής της ομάδος εδώ και επομένως ε, θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησαν οι συνάδελφοι. Το CDM υπήρξε μία μακρά και δύσκολη διαδικασία για επί 12 <coughs> χρόνια. Η Κομισιόν το είπε άλλωστε προηγουμένως. Είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ε, στην ε, μερικές φορές η Ρουμανία ήταν πολύ ευτυχισμένη, άλλες φορές η Βουλγαρία ευτυχισμένη, άλλες φορές και οι δύο ε, απεσιόδοξες. Εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε, ελπίζουμε ότι φέτος ή του χρόνου μέχρι το τέλος τα πράγματα θα έχουν ομολοποιηθεί. Υπάρχει ένα συμπέρασμα από όλα αυτά, τουλάχιστον που εγώ θα ήθελα να εξάγω από όλη αυτή τη διαδικασία. Το είπα και σε προηγουμένως, δηλαδή ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτή η διαδικασία να γίνει ε, κάτι βιώσιμο το οποίο μπορεί πραγματικά να ενταχθεί ε, ουσιαστικά ε, στο κράτος δικαίου. Αυτό που ζητούμε δηλαδή από καιρό και ευελπιστούμε αυτό να γίνει αρκετά σύντομα. Χρειαζόμαστε πανευρωπαϊκό μηχανισμό, εγκάρσιο μηχανισμό ε, κράτος δικαίου, ένα πρότυπο το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί ομοιογενώς σε όλες τις χώρες με σαφείς συστάσεις, με σαφείς ε, επιπτώσεις. Και ε, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, το, ο μηχανισμός ε, συνεργασίας και υποστήριξης δεν θα ήταν απαραίτητος για αυτές τις δύο χώρες. Τώρα όσον αφορά το δεσμό μεταξύ του μηχανισμού CVM και ε, του Σέγγεν, εάν είναι καθαρός, φανερός ή κρυφός και υπόγειος, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι εάν ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και θα προχωρήσουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις και όσο γίνεται πιο γρήγορα να ενταχθεί η διαδικασία ε, monitoring και αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι η σειρά τη κύρια Στράικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς ε, Κομισιόν για τα όσα ε, μας ε, είπατε για τις, την εκτίμησή σας για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Βεβαίω θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ των συντονιστών εάν ε, θα κάνουμε δικιά μας αξιολόγηση, αλλά ε, πράγματι ήδη είναι πολύ ε, ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και μας δίνουν πολλές πληροφορίες. Θα πρέπει να συνεχίσει η αξιολόγηση της Ρουμανίας γιατί έχουμε δει κάποια οπισθοδρόμηση. Από την άλλη μεριά πραγματικά συμμερίζομαι και εγώ τους προβληματισμούς του συναδέλφου που μόλις μίλησε, δηλαδή πόσο αποτελεσματικό πραγματικά ε, ε, αποτελεσματικέ είναι αυτές οι αξιολογήσεις ε, από τη στιγμή που έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Και η δικιά μας ερώτηση είναι η εξή. Τι διδάγματα, τι μαθήματα μπορούμε να αποκομίσουμε από το, την χρήση αυτού του μηχανισμού. τι είναι θετικό, τι όχι, τι μπορεί να ενδυναμωθεί σε αυτό το νέο μηχανισμό. Και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το CDM ε, από τη διαδικασία Σέγγεν. Ε, οι πράσινοι αυτή τη θέση έχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στα απλά μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση που μα παρουσιάσετε λοιπόν εδώ. Και να συγχαρώ την ε, Βουλγαρία για την ε, πρόοδο που πετύχε. Εκ παραλληλού. Είναι τρία χρόνια τώρα που οι Ρουμάνοι έχουν βγει στους δρόμους για να διαδηλώσουν για τα προβλήματα που μαστίζουν την ρουμανική κοινωνία λόγω της κυβέρνησης. Ε. Η, κυβέρ... η έκθεση λοιπόν περιλαμβάνει πολλά στοιχεία τα οποία δεν είναι ιδιαίτερως ακριβή. Το Βουκουρέστι όμως έχει μια καινούργια κυβέρνηση και που έχει δεσμευτεί να σεβαστεί τις συστάσεις του μηχανισμού. και προφανώς θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και τα πορίσματα της Επιτροπής της Βενετίας. Όπως οι συνάδελφοί μου τόνισαν, η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν είναι απόλυτος ενσωματωμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο δεν συμμετέχουν στη ζώνη Σέγγεν. Και θυμάμαι ότι ο υπουργό ε, Μας αναφέραν παραδείγματα και υποδείγματα χωρών ε, ως ε, υποδειγματικές χώρες για το Σέγγεν. Πραγματικά όμως μπορούμε να βάλουμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ του μηχανισμού ελέγχου και συνεργασίας ε, και της ζώνης ε, Σέγγεν. Όλος ο κόσμος το αρνείται αυτό, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Από την Κουέ να ακούσουμε την κυρία Ντάλη. Ναι, είμαι αντίθετη στην ιδέα να κατηγοροποιούνται τα κράτη ως λειτουργικά ή ως μη λειτουργικά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό για διάφορες χώρες. Μιας και συζητήσω όμως, μιας και συζητάμε την Βουλγαρία και τη Ρουμανία, θα περιοριστώ σε αυτές και θα ήθελα να υποβάλω μια μικρή ένσταση σε ό,τι αφορά τη σταθερή πρόοδο που αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την προστασία των μέσων ε, ενημέρωσης και των δημοσιογράφων. Ε, θα ξέρετε ότι οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα αναφέρουν ότι υπάρχουν απειλές και πλέον προειδοποιούν ότι είναι επικίνδυνη η επικράτεια αυτή για τις ανεξάρτητες πηγές ε, ειδήσεων και για την παρενόχληση σε ό,τι αφορά και θέματα υποβολής ερωτήσεων για διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων. Δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις που κατηγορηποιούνται ως ε, επιδοτήσεις για την ελίτ των αγροτών και για μια ελίτ που ε, ωφελείται. Γιατί 75% των ε, αγροτικών επιδοτήσεων δίνεται στη Βουλγαρία και κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί και εμάς στην επικράτειά μου. Στην ε, Πόμερη στην ε, Βουλγαρία ε, έχουν ε, μπει πολλά χρήματα και αυτό ο σκοπό έχει την παράνομη εκμετάλλευση των χρημάτων των ατόμων αυτών με παράνομη χρήση των, του ηλεκτρισμού και του νερού γιατί ουσιαστικά δεν επιτρέπουν στους πόρους αυτούς να χρησιμοποιούνται από άλλους και έτσι δεν ε, μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιήσει και ο κόσμος έχει προσφύγει στα δικαστήρια. Αυτή η εταιρεία ουσιαστικά αλλάζει όνομα κάθε τρεις και λίγο και μετακινείται. Και δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί σε ένα άλλο κράτος μέλλον. Εγώ ως καινούρια βουλευτής, ε, τι μπορώ να κάνω, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσω τους ανθρώπους αυτό, γιατί είναι παράνομο αυτό που συμβαίνει και αποτελεί ντροπή. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Γιόνσεβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ την άρση του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελλάδα και τη Βουλγαρία και ελπίζω να έρθουν και τα εμπόδια για την προσχώρηση της Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν. Έχει δικαίωμα η Βουλγαρία να ανήκει στο χώρο του Σέγγεν. Γιατί κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε όλα τα κριτήρια και να ενταχθούμε σε όλες τις δομές. Δεν θα υπάρχουν πλέον δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι δημοκρατικές αρχές και αξίες δεν μπορούν να γίνονται σεβαστές η δε εφαρμογή αυτών να γίνεται μόνο με ένα εργαλείο, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Θέλουμε και εμείς ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση του κράτους δικαίου. Είμαστε στην πρώτη θέση ε, για την διαφθορά. Επιδεινώνεται η κατάσταση, όπως ε, αποδεικνύει και έρευνα της υπηρεσίας ε, έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου, η PRS. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την διαφθορά, ε, να δείξουμε αποτελέσματα. Δεν τα έχουμε δείξει. Η ετήσια έκθεση της ε, Transparency International δείχνει ότι ξεκολουθούμε μέσα στην πρώτη θέση και σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ η ανεξάρτηση των ΜΜΕ δεν καλύπτεται από το μηχανισμό, επηρεάζει όμως την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Και η δικαστική εξουσία επίσης ε, πλήττεται τα τελευταία δέκα χρόνια εκεί σε ό,τι αφορά την δική μας την κατάταξη. Ήμασταν πριν από κάποια χρόνια στη θέση 34 και έχουμε κατρακυλήσει θέση 111. Αλλά να επαναλάβω, η Βουλγαρία δεν πρέπει να τιμωρείται λόγω των πολιτικών που έχει, αλλά πρέπει να ενταχθεί πλήρως στη ζώνη Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Βιτάνοφ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βουλγαρία είναι θετική και θέλω να υπογραμμίσω εδώ πως ε, όλοι μας, ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας, Κάναμε πολλές προσπάθειες ώστε να πάψει να ισχύει πλέον ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου. Ήταν άλλωστε μια απλή διατύπωση τα τελευταία χρόνια. και οι εκθέσεις χρησιμοποιούνταν ως όπλο για τις εκλογές. Δεν ήταν ένα απλό τεχνικό εργαλείο. Έγιναν δηλαδή πολιτικό εργαλείο. Ε, χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ε, η όλη κατάσταση ε, και σε ό,τι αφορά τις την πρόοδο που σημειώνει η χώρα. Όλα αυτά τα εκμεταλλεύονταν στι εκστρατείε πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Um, Εσείς, ε, κύριε Τσιχουντάρου, ελπίζω να το είπα σωστά το όνομά σα. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρουμε τους βουλγαρούς φίλους για την επιτυχία τους. Πρέπει να έχουμε όλοι όμως την ίδια μεταχείριση είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θεσπίστηκε το 2007 κατά, ε, κατόπιν δικού μας αιτήματο. Ήταν ε, τεχνικό το μέτρο, όχι, ήταν ένα οργανωτικό μέτρο από το 2009. χρησιμοποιήθηκε σε μας και είπαμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση για όλους. Είναι τελείως λάθος η βάση που εδράζεται. Τι προεξόφλημα αποτέλεσμα. Όλο και περισσότεροι λένε ότι τα δεδομένα σε εκθέσεις αυτές είναι ψευδή ή εσφαλμένα. Και πρέπει να τις ξαναεξετάσουμε όλες αυτές τις εκθέσεις. Στο Σύνταγμα μιλάμε στη χώρα μου για ισότητα μεταχείριση όλων ίσως ο νέος μηχανισμός ε, παρακολούθησης για το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη να ήταν η λύση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και ελπίζουμε να πετύχει αυτή η νέα προσέγγιση. Όλοι έπρεπε να είναι αντικείμενο αυτού του μηχανισμού. Πότε λοιπόν θα τεθεί σε αυτός ο μηχανισμός. Θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να ευκρινίσω. Και καλό είναι να ακουστούν στα αγγλικά. Ακούσαμε, την, διάβασα την έκθεση και την πολιτική και την τεχνική για τη Ρουμανία με μεγάλη προσοχή. Πριν εκλεγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπούσα μία μικρή από τη ΣΥΠΑ, η οποία για πολλά χρόνια πολεμούσε την καταπολέμηση της, για την καταπολέμηση της ε, διαφθορά στη Ρουμανία και για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους, για όλους τους Ρουμάνους. Επί σειρά ετών, λοιπόν, υπήρχαν ε, πολύ βασικέ ε, παραβιάσει των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων των Ρουμάνων και διάβαζα λοιπόν την έκθεσή σα και θα ήθελα να υποδείξω κάποια τεχνικά ασφάλματα, κάποια ποσοτικά ασφάλματα, κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν βάση που μα κάνουν και ανησυχούμε για την αντικειμενικότητα τη έκθεση σα. Κάποια παραδείγματα. Σε μια υποσημείωση αναφέρεται το εξή. Το Νοέμβριο του 2018 2.300 ε, περιπτώσεις είχαν να κάνουν με δικαστές που είχαν καταχωριστεί μεταξύ του 1940 και 2000. Αυτό είναι λάθος και δεν στέκει. Στην περίοδο αυτή είχαμε 2.901 περιπτώσεις δικαστών. Αυτός ο αριθμός μπορεί να σημαίνει κάτι για κάποιους και να μην σημαίνει τίποτα για κάποιους άλλους. Είχαμε 7.000 δικαστές στην ε, Ρουμανία. Αν δείτε λοιπόν τα ποσοστά πάνω από το 40% των ε, δικαστών μεταξύ 2014-2018 είχαν ξεκινήσει ε, υποθέσεις και καταπολέμηση διαφθοράς. Οι ειδικέ λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες στη Ρουμανία έχουν να κάνουν ε, με συγκεκριμένες με ε, ατασταλίες από κάποια ομάδα και όχι από όλες τις ομάδες. Και αυτό δεν στέκει. Το γεγονός ότι, ε, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι αυτά είναι αφιερωμένα μόνο στο στρατό. Αν αναφέρουμε λοιπόν ότι πρόκειται για ανάλυση αλλαγών στην νομοθεσία, τέτοια απλά θέματα δεν στέκουν. Προφανώς. Ο κόσμος στη Ρουμανία και εγώ αναρωτιόμαστε για την αντικειμενικότητα της έκθεσης αυτής. Πέρα από αυτές τις σοβαρές ε, ε, κατηγορία στην έκθεση αυτή, κάτι που μας ανησυχεί και εμάς και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτή αγνοεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαστηρίου και βλέπουμε τι συμβαίνει σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορες ομάδες ανθρώπων και περιφέρειες αρχίζουν, αρχίζουν να αγνοούν τις αποφάσεις του δικαστηρίου, του συντάγματος μάλλον. Ε, αυτά που ορίζει το Σύνταγμα κάποιων χωρών. Αν αρχίσουμε και θέτουμε τέτοια προηγούμενα, πού θα καταλήξουμε οποιοδήποτε μπορεί να αναιρεί και να αμφισβητεί τις αποφάσεις του Σταγματικού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ κύριος Μπούρεκ. Thank you, Mr. Chair. Κυρία Σπούρεκ, ο μηχανισμός ε, για την Ρουμανία και τη Βουλγαρία σχεδιάστηκε ως μεταβατικό μέτρο. Τώρα, με την πρόταση λήξης του CVR για την ε, Βουλγαρία και με την ε, πρόταση ενδυνάμωσης ε, για την άλλη χώρα, μπορείτε να πείτε ότι όλες οι χώρες μέλη στο μέλλον θα υφίστανται την ίδια διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματός τους. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κύριος ε, Πιστεύουμε ότι το κράτος δικαίου και οι μηχανισμοί του θα πρέπει να ελέγχονται και να επιβεβαιώνονται παντού ε, σε όλες τις χώρες και όχι μονάχα στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία παρόν μηχανισμός είναι ένας ε, μηχανισμός ο οποίος αφορά μονάχα δύο χώρες και επομένως δεν είναι συνολικός, ε, κυρίως δεν λαμβάνοντας υπόψη και τα ε, μέσα, μέτρα τα οποία περιλαμβάνει. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα παρακολουθεί το κράτος ε, δικαίου, καθώς επίσης και οτιδήποτε από αυτό απορρέει και επηρεάζει τις δημοκρατικές αρχές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής ε, μηχανισμός προστασίας του κράτους ε, δικαίου που θα καταδεικνύει σε πραγματικό χρόνο που και πότε υπάρχει παραβίαση συγκεκριμένων αρχών και να σημειώνει αυτές τις παραλήψεις οι παραβιάσεις και θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην Ανατολική και την Δυτική Ευρώπη και να λύσουμε τα ζητήματά μας δημοκρατικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, προσυπογράφω ε, τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, σχετικά με την απολύτως ικανοποιητική πρόοδο της ε, Βουλγαρίας ε, και ότι το συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσει που είχε αναλάβει η Βουλγαρία τη στιγμή που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, καλυφθεί. Ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, καταπολέμηση της διαφθοράς σε περιφερειακό και ε, εθνικό επίπεδο και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτά είναι πολύ σημαντικά προβλήματα και παιδεία στα οποία η έκθεση αναγνωρίζει ότι έχει υπάρξει ε, πρόοδος ε, και όσον αφορά τις δικαστικές αρχές και όσον αφορά τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Ωστόσο δεν πρέπει να υπάρχουν διπλά στάνταρ, διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Εδώ και 12 χρόνια ε, υπάρχει ο μηχανισμός αυτός και προετοιμαζόμαστε ε, για μία ε, θετική κατάληξη. Ωστόσο πρέπει να πω ότι πολλές είναι οι χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα με το κράτος δικαίου, με την διαφθορά και επομένως πιστεύουμε ότι ε, θα έπρεπε να υπάρχει ένα είδος μηχανισμού παρακολούθησης για όλους. Μιλισμονούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ε, για συχνές εκθέσεις και αναφορές για την κατάσταση του κράτους δικαίου ε, σε όλες τις χώρες. Και τώρα περιμένουμε βέβαια στην Βουλγαρία την επί τα επίσημα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσει να απαντήσει. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Να ευχαριστήσω και όλους όσους ε, έλαβαν το λόγο για τα σχόλιά τους. Ε, θα σχολιάσω ορισμένα από όσα υπόθηκαν για, τη για το ζώνη Σέγγεν καταρχάς. Είμαστε συνεπείς στην Κομισιόν στην προσέγγιση και στην άποψή μας ότι δηλαδή είναι λάθος να γίνει ε, διασύνδεση μεταξύ του μηχανισμού συνεργασίας και έλεγχο και του Σέγγεν αφετέρου αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Για τις ερωτήσεις που ακούστηκα σε σχέση με τη διαδικασία. Πώς ξεκίνησε ο μηχανισμός το ξέρουμε. Ουσιαστικά βασίστηκε στη δέσμευση για προσχώρηση. Είναι ιστορικό το θέμα και όσο ό,τι αφορά τη διαδικασία. Κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται και η Κομισιόν θεωρούμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. η δουλειά μας έχει ανατεθεί. Θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, να ακούσουμε όλες τις πλευρές, να ελέγξουμε όλες τις λεπτομέρειες. Και επίσης οι αρχές των δύο κρατών μελών επίσης μελετούν το κείμενο για να ελέγξουν τα γεγονότα, τα, το κατά πόσο μεταφέρονται όλα σωστά κτλ. Η διαδικασία αυτή ήταν. Και πάντοτε ε, ήταν ε, θετικά τα σχόλια του Συμβουλίου στα συμπεράσματά του για τη διαδικασία. Και τα συμπεράσματα συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτό που θα έλεγε κανείς διεθνή συνένεση για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Επιτροπή της Βενετίας και άλλους ε, εξέχοντες φορείς αντίστοιχους για την ερεσιμότητα. Η έκθεση για τη Ρουμανία δεν νομίζω ότι θα ζητήσει καθέναν τρόπο ε, το σύνταγμα. Συνταγματικότητα, πολιτική δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί κανείς να είναι συνταγματικός αλλά να μην κάνεις ε, τη σωστή πολιτική κατά την άποψη τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Δηλαδή ότι δεν ευθυγραμμίζονται οι πολιτικές πάντοτε με του επιδιωκόμενου στόχους. Σε ό,τι αφορά τώρα τι μεμονωμένε περιπτώσεις, ο μηχανισμός συνεργασία και ελέγχου έχει να κάνει κυρίως με συστημικά ζητήματα, ενώ για τις μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί. παραδείγματο χάρη για την κατάχρηση κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και φυσικά υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα μας προσφέρει ένα ακόμη εργαλείο για να σημειώσουμε πρόοδο στους τομείς αυτούς. Πιστεύω ότι ένα θέμα πολύ σημαντικό, όπως φάνηκε από τα ερωτήματα, είναι η μετάβαση σε ένα σύστημα δηλαδή που θα αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης όρις, σύστημα παρακολούθησης κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Αν δείτε τι προτείνουμε για τη Βουλγαρία, είναι δύο ουσιαστικά τα στοιχεία. Πρώτον, η πλήρωση των ε, υποχρεώσεων ή τέλο πάντων ε, εφαρμογή των συστάσεων και δεύτερον, δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος με τον νέο μηχανισμό κράτους δικαίου. Αυτό το τονίσαμε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές ξεκάθαρα διαστόματος της, προέδρου, ε, της νέας Προέδρου της Κομισιόν. Η Κομισιόν πραγματικά θα επιδιώξει την θέσπιση αυτού του μηχανισμού. Σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης όρις. Και νομίζω ότι έχουμε αντλήσει διδάγματα από το μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου. Για να δούμε πώς μπορούμε να καταρτήσουμε αυτό το νέο σύστημα που θα βάζει σε ίδιο επίπεδο όλα τα κράτη-μέλη που θα λαμβάνει υπόψη και κάποιες παραμέτρους που υπάρχουν και στο CVM. Υπάρχουν βέβαια κάποιες παράμετροι που δεν λαμβάνονται υπόψη στο CV, όπως είναι τα ΜΜΕ. Εμείς θέλουμε να έχουμε στο μέλλον μια ισότιμη βάση για όλους, αλλά να μπορούμε να εξετάζουμε και το πλήρες φάσμα του κράτους δικαίου. Επεκτείνοντας το πεδίο του CVM. Και αν δούμε μπροστά, Έχετε η Ρουμανία αυτά τα δύο στοιχεία, το νέο περιβάλλον και τις συστάσεις. Αυτό δείχνει ποιο είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε για να ε, πάψει να ισχύει στην περίπτωση της χώρας σας ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέρες θέλει ξανά το λόγο. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Μου προκάλεσε μεγάλη, μεγάλο σοκ αυτά που είπατε. Ότι είπατε ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι συνταγματικά, αλλά να μην συνάδουν με την ε, πολιτική. Με την πολιτική πιανού. Όλες οι δημοκρατίες ε, στην Ευρώπη είναι ε, συνταγματικές δημοκρατίες. Όταν έχει κανείς πρόβλημα, πηγαίνει στο δικαστήριο, πηγαίνει στο συνταγματικό δικαστήριο και Υπάρχουν και οι δύο πλευρές και οι δύο συμβαλόμενοι ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο λοιπόν εισακούει και τις δύο πλευρές και αποφασίζει, αποφαίνεται. Αυτό που αναφέρεται και το προηγούμενο που θέτεται και είχα δίκιο όταν το υπογράμμισα αυτό. Οποιαδήποτε χώρα λοιπόν θεωρεί τι, ότι μπορεί να υπονομευθεί να η δημοκρατία κάθε χώρας από κάποιον ο οποίος ε, επικαλείται μια πολιτική υπονομεύει το Σύνταγμα της χώρας. Μία ερώτηση λοιπόν έχω να κάνω. Ποιος την έγραψε αυτή την έκθεση για τη Ρουμανία, ποιος είναι ο εμπειρογνώμονας και ποια είναι η τεχνογνωσία αυτών των ανθρώπων στην τελική ανάλυση. Να είμαι σαφής από αυτού για το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης των συνταγματικών δικαστηρίων. Αυτά καθορίζουν τα συνταγματικά ζητήματα. Αλλά κοιτώντα τους ε, νόμους και τις πολιτικές. Υπάρχουν συνταγματικά ζητήματα και υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν είναι συνταγματικά. Επιλογές πολιτικής, για παράδειγμα, αυτά τα θέματα επισημαίνει και εξετάζει η έκθεση, όχι τα συνταγματικά ζητήματα. Είναι διαφορετικά ζητήματα, λοιπόν. Τώρα, σε σχέση με το Ποιο κατάρτισε την έκθεση, θα ήθελα να σας πω ότι κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια θέματα και η απάντηση είναι η ίδια. Αυτά τα επιβεβαιώνει και το Συμβούλιο όλων των κρατών μελών. Όλα τα κάτι μέλη έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Έχει εγκριθεί αυτό από το σώματων της Επιτροπής και αποτελεί έγγραφο επίσημο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το θέμα αυτό και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη. Преминаваме 24. και να περάσουμε στο σημείο 24 τώρα για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επαλήθευση της πλήρους εφαρμογής του κεκτημένου Σέγγεν από την Κροατία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ακούσουμε μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ανακοίνωση 11 Οκτωβρίου του φετινού έτου για την επαλήθευση τη πληρού εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν από την Κροατία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στου αντιπροσώπους ε, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν θέλουν να πάρουν το λόγο μετά και οι βουλευτές. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Good afternoon. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα κύριε και κύριοι και αγαπητοί βουλευτές. Το 2015 η Κροατία δήλωσε την προθυμία της να ξεκινήσει την διαδικασία εξελόγησης Σέγγεν σε όλους τους σχετικούς τομείς. Μετά από την δήλωση αυτή προθυμίας της Κροατίας, η διαδικασία για το Σέγγεν ξεκίνησε το 2016. Μέχρι τα μέσα του 2019 η αξιολόγηση Στου τομεί τη προστασία δεδομένων, συνεργασία, αστυνομική, πολιτική για τι θεωρήσει ε, σύστημα πληροφόρησης, σε ό,τι αφορά τα όπλα και σε ό,τι αφορά την δικαστική συνεργασία, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ειδοποίησε σχετικά την Κροατία. Να κοιτάξουμε το θέμα των εξωτερικών συνόρων, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο μεγαλύτερου ελέγχου στην διαδικασία ελέγχου Σέγγεν. Η πρώτη αξιολόγηση έλαβε χώρα, μάλλον η πρώτη αποστολή έλαβε χώρα το Μάιο του 2016. Μετά από αυτό ακολούθησαν δύο επισκέψεις, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2017 και τον Μάιο του 2019. Οι πρώτε δύο επισκέψει έλαβαν χώρα το 2016 και το 2017 και κατέληξαν σε πορίσματα μη συμμορφώσει ή τρίτη επίσκεψη το 2019 κατέληξε σε πορίσματα συμμόρφωσης ε, που επιδέχονται όμως βελτίωσης. Την τελευταία επίσκεψη το Μάιο του 2019 επιβεβαιώθηκε επίσης ότι κάποιες από τις συστάσεις στις προηγούμενες επισκέψεις ε, έπρεπε να εφαρμοστούν. Το σχέδιο του κανονισμού το Μάιο μάλλον της επίσκεψης για το Μάιο του 2019 έλαβε θετικές αντιδράσεις από όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην Επιτροπή Σέγγεν στις 5 Σεπτεμβρίου του 2019. Εν τω μεταξύ και μετά τα συμπεράσματα τα οποία εξαγάγαμε στην επίσκεψη του 2019 η Κροατία εμ, έδωσε εκθέσεις follow-up προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των συστάσεων σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις του 2016 και 2017 και περαιτέρω διευκρινήσεις το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και τον Μάιο και τον Ιούλιο. Υπήρχε δηλαδή ουσιαστικά μηνιαία υποβολή εκθέσεων από πλευρά της Κροατίας, η οποία καταδείξε σημαντική πρόοδο. Και να κοιτάξουμε λίγο πιο πολλές λεπτομέρειες για τα θέματα των συνόρων ένα ζήτημα το οποίο ε, επιτέχεται περαιτέρω διευκρινήσεις είχε να κάνει με το προσωπικό των συνοριοφυλάκων. Κατά την ετήσια υποβολή εκτέσεων, διευκρινίστηκε ότι το προσωπικό της συνοριοφυλακής και των χερσαίων συνόρων και τον αρχικό σχεδιασμό, ε, τήρησε τον αρχικό σχεδιασμό της Κροατίας. Να έχουμε επίσης υπόψη μας ότι μόνο μόλις σταματήσουν οι εσωτερικοί έλεγχοι θα μπορέσουν να μετακυριθούν ε, συνοριοφύλακες από τα σύνορα με τη Σλοβενία και την ε, προς τα εξωτερικά σύνορα με την Σερβία την Μαυτοβραβούνιο. Και Είχαν γεννήσει επίσης συστάσεις το Μάιο για την ανάγκη να αναβαθμιστούν οι δυνατότητε για την ε, επιτήρηση των χερσαίων συνόρων. Εδώ, ενώ όλα τα στοιχεία υπήρχαν πλέον, για να υπάρχει καλύτερη σχέση μεταξύ των τεχνικών ικανοτήτων που έχει η Κροατία και του προσωπικού σε ό,τι αφορά και την ανάλυση κινδύνου. Ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε. Αυτό πλέον ως αρχή είχε εφαρμοστεί από την Κροατία. Αυτό φάνηκε από τις αιτήσεις εκθέσεις. Άλλα θέματα όπου η Κροατία σημείωσε καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά την τεχνική παρακολούθηση στα εξωτερικά σύνορα με την Βοσνία, Ζεγοβίνη και με το Μαυροβούνιο η Κροατία κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία για τις δημόσιες συμβάσεις για τα κινητά τέτοια οχήματα. Στην σελίδα 6 λοιπόν των συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι μετά από αξιολόγηση της πρόοδου που σημείωσε η Κροατία μετά την επίσκεψη του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Κροατία πλέον έχει λάβει τα μέτρα που χρειάζεται για να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για τη ζώνη Σέγγεν και για την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Η Κροατία θα συνεχίσει να... θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή για να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι αυτοί. Άρα, θα πρέπει να γίνει ακόμα κάποια δουλειά σε ό,τι αφορά την κανονική διαδικασία αξιολόγησης ε, Σέγγεν. Από την άλλη, η Κροατία έχει λάβει όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Τετραετής λοιπόν ε, περίοδος ε, παρακολούθησης κατά, τις οποίες, κατά την οποία η Κροατία έκανε τις δέουσες προσπάθειες για να συμμορφωθεί. Και γι' αυτό λοιπόν στη σελίδα 14 στο τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεραίνει όχι μόνο για τα εξωτερικά σύνορα, αλλά και για όλο το συγκεκριμένο Σέγγεν, ότι η Κροατία έχει λάβει τα μέτρα που χρειάζονται για να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι. Ότι η Κροατία θα συνεχίσει. Θα πρέπει να συνεχίσει να προβαίνει προς τις σχετικές ε, ενέργειες και θα καλέσουμε τώρα το Συμβούλιο να εγκρίνει την ανακοίνωση αυτή και να περάσει στα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τους συντονιστές, την κυρία Ματσόλα πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτήν την ε, πολύ αναλυτική παρουσίαση του θέματος. Θα είμαι σύντομη. Ε, η έννοια της, ε, του Σέγγεν, ε, ε, κυρίως σε σχέση με τα εξωτερικά σύνορα, είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική και πρέπει να είναι αυστηρή. Μετά από πολλές προσπάθειες που κατεβλήθησαν από πλευρά της κρατικής κυβερνήσεως, είναι έτοιμοι να ενταχθούν στον χώρο Σέγγεν και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι η παρουσία της Κροατίας στο χώρο Σέγγεν θα ενισχύσει την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο κύριος Τσιριτάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, λέγομαι ε, Τσούχο Νταρού και είμαι ε, γιατρός στα κατεπήγοντα, στο τμήμα κατεπηγόντων ενός νοσοκομείου στην Τιμισοάρα. Θα επαναλαμβάνω το όνομά μου μέχρι να το μάθετε απ' έξω. Αγαπητοί Κομισιόν, δεν μπορώ να μην μιλήσω για τα προβλήματα τα οποία ισχύουν και για την Ρουμανία. Ε, πότε θα μπει η Ρουμανία επιτέλους στο χώρο Σέγγεν? Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω, λέει ο Πρόεδρος, να υπάρχει κάποιο από το Ρενιού. Επομένως, η κυρία Στράικ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ιδιαίτερα σε ευχαριστούμε την Κομισιόν για την παρουσίαση και την έκθεση. Θα ήθελα να εστιάσω στο θέμα το, της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων ε, σε σχέση με ε, τα σε σχέση κυρίως με την διαδικασία ασύλου εγώ έκανα μία ε, μελέτη όσον αφορά τα pushbacks, τις επαναπροωθήσεις ε, και μελέτησα επίσης ε, ε, και κατηγορίες ε, από, τις, ε, από την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τον διαμεσολαβητή, τον συνήγορο, τον ομπουτσμαν της Κροατίας. Δηλαδή είναι, θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται εάν καταφέρνουν κάποιοι να περάσουν τα σύνορα, εάν επαναπροωθούνται, εάν αφού περάσουν τα σύνορα ξεκινάει μια πραγματική διαδικασία ασύλου κλπ ή εάν έρχονται ε, σε ε, ε, αν έρχονται σε αντιπαράθεση με στρατιώτες του κροατικού στρατού που τους αποθούν και τους επαναπροωθούν. Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν, έχει γίνει αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών. Επίσης, η διατύπωση για μη συμμόρφωση ε, και για ε, τις προκλήσεις που παραμένουν ε, δεν είναι πολύ σαφή για μένα. Αν δείτε το άρθρο 40, αναφέρεται ότι... Όχι, μάλλον έχω κάνει λάθος, λέει ο Μιλήτρια. Αναφέρει ότι η διαδικασία ε, της, ε, του ελέγχου των συνόρων θα πρέπει να παραμείνει πλήρως συμμορφούμενη και αργότερα λέει ότι η Κροατία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Ερώτηση λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Κομισιόν συμπεραίνει, παρατηρεί ότι οι παρούσες πρακτικές ε, όσον αφορά τη διαδικασία ασύλου στις κροατικές αρχές ε, με το τον ε, έλεγχο συνόρων και με τον κώδικα Σέγγεν καθώς επίσης ε, με το κεκτημένο για το άσυλο και με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι σαφή αυτά κατ' μέ Επίσης, ε, νέος monitoring mechanism, μηχανισμός επιτήρησης αναφέρθηκε. Πώς θα λειτουργεί αυτός ο νέος μηχανισμός επιτήρησης, θα υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Επίσης, πώς μπορούμε να επιτηρήσουμε αυτήν την κατάσταση, κυρίως όσον αφορά τις επαναπροωθήσεις. Η κεντρική μου ερώτηση είναι ε, υπάρχει συμμόρφωση και με ποιο τρόπο και αν δεν υπάρχει συμμόρφωση πώς ξέρουμε ή πώς περιμένουμε ότι θα προκύψει συμμόρφωση γιατί αυτό είναι πολύ αποφασιστική σημασία κριτήριο ε, πριν αποφασίσουμε ε, την... Ε, πρόσβαση στο Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάλη από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις, λίγος χρόνος. Πάντα αυτό συμβαίνει. really in the of... Άκουσα προσεκτικά τη δήλωση της, ε, προσοχή, της ε, Κομισιόν, αλλά και εσείς οι ίδιοι λέτε ότι παρά τα τέσσερα χρόνια και τις διαρκείς παρακολουθήσεις ε, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Εμείς γνωρίζουμε ότι στα, συμφέρο, στα σύνορα της εκρωτίες και της Βορσίας ε, ε, Ζεγοβίνης γίνονται συστηματικά επαναπροωθήσεις και παραβιάσεις. Τι μας λέτε, ότι εάν υπάρχουν χώρες οι οποίες ελέγχουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τότε θα πρέπει να γίνονται μέλη ε, ε, Σέγγεν και παρά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις διαδικασίας ασύλου κλπ. Ε, δηλαδή ε, μιλάμε με μεγάλο ενθουσιασμό για τη διαχείριση των συνόρων και την προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά μετά όλη αυτή η ιστορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο βαρετή πώς, πώς ε, επίσης ε, και σε σχέση με τις νέες εξελίξεις, ε, πώς θα δώσει η Κομισιόν το πράσινο φως, ποια θα είναι η θέση του Κοινοβουλίου, ποιες οι δυνατότητες να παρέμβει, γιατί υπάρχουν και κάποια νομικά ζητήματα τα οποία είναι πιο σημαντικά από, τη, από άλλα αλλά όλα τα κριτήρια του Σέγγεν νομικώς θα πρέπει να καλύπτονται. Αυτό όμως δεν συμβαίνει εδώ. Ε, και εξειδικευμένα χρειαζόμαστε απαντήσεις ε, ε, σχετικά με το ποιες δράσεις ελήφθησαν υπόψη όταν μελετήθηκε η συμμόρφωση της Κροατίας προς το άρθρο 4 του κώδικα Σέγγεν όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχουν στοιχεία για τα οποία δεν έχει απαντήσει ακόμα η κροατική κυβέρνηση όσον αφορά το σχέδιο δράσης θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, βελτιωθούν ε, ε, οι καταστάσεις όπου ξέρουμε ότι είναι προβληματικές αλλά πώς είναι δυνατόν να δώσουμε το πράσινο φως πρώτα θα απαντηθούν τα ερωτήματα πρώτα θα λυθούν τα προβλήματα και μετά θα προχωρήσουμε Σας ευχαριστώ Κύριε Ρέστλερ Ευχαριστώ να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για να μπορούν οι Κροάτες υπηκόοι να απολαμβάνουν ε, μία από τις μεγαλύτερες ε, επιτυχίες της Ένωσης που είναι ελευθερία κυκλοφορίας πρέπει η χώρα να εκπληρώσει τα αυστηρά κριτήρια προσχώρησης ε, στη ζώνη του Σέγγεν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί από ΜΚΟ και λόγω αυτών και του πλαισίου γενικώ χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τώρα η μόνη αρμόδια αρχή η οποία πραγματικά μπορεί αντικειμενικά να αξιολογήσει τεχνικά την κατάσταση, επιβεβαιώνει ότι η Κροατία πληρώνει πλέον, εκπληρώνει όλα τα αυστηρά κριτήρια και μπορεί να προσχωρήσει. Πάνω από 6.000 κράτε αστυνομικοί σήμερα προστατεύουν ε, τα πιο μακρά σύνορα της Ένωσης. Χαιρόμαστε που με την προσχώρηση της Κροατίας θα έχουμε καλύτερες συνδέσεις, οικονομική συνεργασία, έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Και για όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι προς το συμφέρον όχι μόνο της Κροατίας αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσχώρηση της Κροατίας στη ζώνη Σέγγεν. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. σας ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Μαρκουάρτ. αν δεν έχετε πρόβλημα, λέει ο κ. Μαρκάτ, να τα πω στα γερμανικά. Και εγώ νομίζω ότι είναι προ το συμφέρον και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο και των Κροατών η προσχώρηση δηλαδή της ε, Κροατίας στη ζώνη Να Θεωρώ ότι είναι και προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είμαστε ειλικρινεί ε, ο ένας απέναντι στον άλλο. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες από μιμικιό και λέμε ότι είναι υποκειμενικές, ενώ απ' την άλλη υπάρχουν αντικειμενικές απόψεις ε, που λένε ότι όχι αυτά που λένε μικιό δεν συμβαίνουν. Δεν είναι όμως μόνο οι μικιό που τα λένε και εγώ έχω πάει στα σύνορα, έχω μιλήσει με κόσμο εκεί και πραγματικά ε, είναι προφανές ότι αυτά τα βίντεο ε, έχουν ε, γίνει προφανώς από άτομα τα οποία τα βλέπει κανείς εκεί και στα σύνορα με τη Βοσνία ότι τους έχουν καταστρέψει τα κινητά, έχουν σπασμένα κόκαλα, έχουν πληγές και σημάδια και τους σπάσαν τα κινητά τους και δεν ξέρω εγώ τι και τους ε, προσπαθούν να εκφοβήσουν να πάνε στην Κροατία. Στην ε, Κροατία συστηματικά ε, τους αρνούνται σε αυτούς τους ανθρώπους να τους ε, χορηγηθεί άσυλο και τους αποθούν. Επομένως δεν είναι απλά κάποιες καταγγελίες ή ισχυρισμοί ε, ανυπόστατοι που κάποιος τους έχει έτσι εφεύρει, αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Λέμε ότι είναι προς το συμφέρον ε, της Κροατίας και των Κροατών να είναι μέλος ε, του Σέγγεν. Τότε είναι προς το συμφέρον μας να εκπληρεί η χώρα όλα τα κριτήρια και όχι επειδή είναι έτσι η κατάσταση, γιατί ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση. Λένε κάποιοι ότι αυτή η κατάσταση που εγώ σας περιέγραψα δεν υπάρχει. Άλλοι όμως που είναι επιτόπου λένε κάτι τέλος διαφορετικό. Πρέπει να υπάρξει ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη Πώ θα οικοδομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη, Πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό το πρόβλημα στην Κροατία. Υπάρχουν παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι μια σοβαρή παραβίαση, είναι σοβαρό πρόβλημα. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την κατάσταση, τώρα πώς την περιγράφουν. Εγώ τα είδα και έχω την προσωπική μου άποψη. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά που λέω εγώ ισχύουν ή υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε από πού θα ξεκινήσω. Να δούμε ένα προς ένα θα τα πιάσω. Λοιπόν, ξεκινώ με τα θεμελιώδη δικαιώματα ένα από τα μείζωνα ή το μείζον ζήτημα που ετέθη. Και τις αποθήσεις συγκεκριμένα θέλω να αναφέρω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέταστο το κατά πόσον έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η Κροατία για την προσχώρησή της στα θέματα των δικαιωμάτων και επιβεβαιώνει στην ανακοίνωση της η Κομισιόν το γεγονός ότι η Κροατία συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο για τη βελτίωση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχουν τώρα, είπαμε, κάποιοι ισχυρισμοί για την μεταχείριση ετούντων άσυλο. Πρέπει να γίνουν έρευνες από τις κρατικές αρχές που θα είναι αξιόπιστες με βάση το διεθνές δίκαιο θέλουμε σύντομα, αμελητή, να ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις η Κροατία και να τηρεί ενήμερη την Κομισιόν. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση. Πρέπει να έχετε επίσης υπόψη ότι όταν εκτεθεί απόφαση επίσημη του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Κροατίας θα μπορεί αυτεπάγγελτα και απροειδοποίητα να κάνει ελέγχους η Κομισιόν. Αλλά προς το παρόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς είναι προγραμματισμένες επισκέψεις, οπότε χάνεται το στοιχείο της έκπληξης, του ευνηδιασμού στα εξωτερικά σύνορα. Αυτές λοιπόν οι απροειδοποίητες επισκέψεις ε, θα μπορούν να γίνονται εφόσον αρθούν οι έλεγχοι στα σύνορα. Και αυτό σίγουρα θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην Κομισιόν. Θα μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο δεν θέλαμε να περιμένουμε τόσο πολύ και γι' αυτό κατόπιν αιτήματος ε, της ε, Κομισιόν ε, θεσπίστηκε μηχανισμός παρακολούθησης με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι συνεργειακές δραστηριότητες στα σύνορα να τηρούν τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και να υπάρχει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει το κεκτημένο ασύλου. Πώ μπορέσαμε να τα ελέγξαμε όλα αυτά, δώσαμε 6,8 εκατομμύρια ευρώ στην Κροατία από το Δεκέμβριο ήδη του 2018 σε κατεπίγουσα επιχορήγηση και υπάρχει αυτός ο μηχανισμός τώρα που έχει ως αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα και η συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ε, ενεργειών στα σύνορα. Τρεις βασικοί στόχοι της παρακολούθησης. Πρώτο και σημαντικότερο παρακολούθηση της συμπεριφοράς των αστυνομικών επιτόπου ε, σε ό,τι αφορά τη λαθρομετανάστευση και την παράτυπη μετανάστευση και του ε, τον τεσάσυλο. Υπό την ΥΠΑΤΗ και το Κέντρο Δικαίου της Κροατίας και υπάρχουν εκπρόσωποι των συνοροφυλάκων ε, και των ε, αρμοδίων υπουργείων του Υπουργείου Εστερικών μεταξύ άλλων. Κάτι άλλο είναι η εκπαίδευση για να αλλάξει νοοτροπία ο κόσμος, να καταλάβει ότι οι μετανάστες, οι άνθρωποι που χρήζουν διεθνούς προστασίας, πρέπει να έχουν μια αξιοπρεπή μεταχείριση, αξιοπρεπή Εκπαίδευση των αστυνομικών λοιπόν η δεύτερη συνιστόσα του μηχανισμού παρακολούθηση για τον οποίο προσπαθώθηκαν 6,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εκπαίδευση και πάλι γίνεται από την υπεταρμοστία για τους πρόσφυγες και από διάφορες οργανώσεις και των πολιτών, αλλά δεν μιλάμε μόνο για εκπαίδευση. Μιλάμε και για τις ε, κανονικές συνήθεις ε, πρακτικές, επιχειρησιακές πρακτικές από τη μεθοριακή αστυνομία ε, και εδώ επαναλαμβάνω συμμετέχει και το κέντρο δικαίου και η πατερμοστία για τους πρόσφυγες. Και το τρίτο στοιχείο είναι η συνεργασία των κρατικών αρχών με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με διάφορα εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτός ο μηχανισμός παρακολούθησης που θεσπίστηκε το Δεκέμβριο της περσινής χρονιάς εξασφαλίζει την ανεξάρτητη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και ενεργειών της μεθοριακής αστυνομίας της Κροατίας. Αυτός ο μηχανισμός παρακολουθησής εν τέλει συμπληρώνεται με ένα πρωτόκολλο του Υπουργείου Στερικών της Κροατίας και της ΕΠΑ και του Κέντρου Δικαίου της Κροατίας για την παρακολούθηση των συνοροφυλάκων αυτών. Η χρηματοδότηση ευρωπαϊκή ήταν ε, πραγματικά κομβική σημασίας για να γίνει πράξη η παρακολούθηση και η εκπαίδευση εκεί, παρότι είναι ένα πιλωτικού προγράμματο. σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, είναι γνωστή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλές φορές το υπογράμμισε και ο ίδιος ο Επίτροπος Αβραμόπουλος. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εκπληρούν τα κριτήρια για την προσχώρησή τους ε, στη ζώνη του Σέγγεν. Και αν τα πληρούν μπορούν να μπουν στο Σέγγεν και να έρθουν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία λοιπόν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και οι δύο χώρες κατά την άποψη της Κομισιόν είναι πλήρως έτοιμες να προσχωρήσουν στο Σέγγεν. Η απόφαση τώρα είναι πολιτική και πρέπει να ληφθεί ομόφωνα από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτά λοιπόν είπα ε, για τις αποθήσεις, τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάλη για ένα λεπτό, ναι. Μια και έχουμε χρόνο και δεν νομίζω ότι ήταν πολύ λεπτομερή η απάντηση για να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Θα ήθελα πιο πολλέ πληροφορίε. Πότε ιδρύθηκε ο μηχανισμό, ο νομισματικό μηχανισμό και σε ό,τι αφορά την υπατή αρμοστία του ΟΗΕ και την κρατική πλευρά παρακολουθεί την κατάσταση. Υπάρχει μια σταθερή ομάδα παρακολούθηση σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Πόσοι αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν, το ξέρετε αυτό. Ποιο επέβλεψε το έργο αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα νομικά λοιπόν ε, κριτήρια δεν πληρούνται ακόμα και παρόλα αυτά μα λέτε ότι η συμμετοχή της Κροατίας στο Σέγγεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό θεωρώ ότι είναι παρόνομα, γιατί όλες οι νομικές διατάξεις είναι ίσες και μας είπατε ότι οι νομικές διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν εκπληρούνται. Πώς λοιπόν δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός παρακολούθησης και τις συγκεκριμένε ημερομηνίες, πότε λάβανε χρήματα κτλ. κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρκαρτ για ένα λεπτό. Για να είμαι σύντομο, δεν ε, θέλω να κατηγορήσω τους ε, μεμονωμένους αστυνομικούς, αλλά από ό,τι ακούω από τις διάφορες ε, πλευρές είναι ότι ήταν τεράστια η πίεση, η πολιτική πίεση στην ε, κρατική αστυνομία, στην φυλακή που αυτό ενδεχομένω να, να σε εγκλήματα. Υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη για τις συνέπειες που ε, αναγκάζονται να υποστούν οι, οι συνοριοφύλακες σε ό,τι αφορά τις επαναπροωθήσεις. Υπήρχαν, ε, για παράδειγμα, συνέπειες για αστυνομικούς που αρνήθηκαν να παραβιάσουν το νόμο. Ευχαριστώ πολύ. Και κύριος Ρέστλε, ένα σχόλιο ακόμα. Ήταν περίπλοκη η νομική και η τεχνική αξιολόγηση. Πήρε πολλούς μήνες και επιβεβαίωσε τις τεχνικές διορθώσεις και βελτιώσεις που έκανε η κρατική αστυνομία και η κρατική κυβέρνηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφύγουμε. Να μην δώσουμε πολιτική διάσταση ε, σε μια έκθεση η οποία ουσιαστικά αποτελεί τεχνική αξιολόγηση και μάλιστα έγινε για ένα, σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στράικ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με το τελευταίο σχόλιο. Δεν θα πρέπει να πάρει πολιτικό χαρακτήρα η συζήτηση. Και το, αυτό που με εντυπωσιάζει είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ των συμπερασμάτων των θεσμικών οργάνων. Ο, διεθνής, ο Εθνικός Διεθνής κτλ. Και τις τάσεις των εθνικών αρχών. Αν όντω είπατε ότι δεν επιτρέπονται οι ευνηδιαστικέ ε, επιθεωρήσει, πώ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και ότι η κατάσταση είναι σχεδόν συμβατή. Άρα, επί ποιας βάσης λάβατε τα... τις αποφάσεις σας. Και επίσης, ο μηχανισμός παρακολούθησης υπάρχει πλέον εδώ και ένα χρόνο. Ποια είναι τα αποτελέσματα, ποια είναι τα απορίσματα... Μπορούν να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα βάσει του μηχανισμού αυτού και πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες βάσει του μηχανισμού παρακολούθησης αυτού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέφερτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Το ε, project ε, ξεκίνησε το 10, Σεπτέμβρη 18, το Σεπτέμβριο του 18 και έχει περίπου ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται σε ένα ε, μήνα. Αυτό δηλαδή για την επίγουσα ε, κατάσταση όσον αφορά τα υπόλοιπα. Ε, μπορώ να σας πω ότι θα υπάρξει μία στρογγυλή τράπεζα ε, όπου θα συζητηθούν τα αποτελέσματα. Οι κροατικές αρχές μας έχουν υποβάλει εκθέσεις ε, προόδου που θα συζητηθούν στην τελική στρογγυλή τράπεζα που θα λάβει χώρα σε, μερικούς εβδομάδες. σε μερικές εβδομάδες. Θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Η Κομισιόν συγχρηματοδότησε το project ε, και η Κροατία ως δικαιούχος οφείλει να υποβάλει η τελική έκθεση στην Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα το θέμα σχετικά με το ποια είναι η άποψη της Κομισιόν Δυστυχώς δεν είμαστε επιτόπου, ε, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί επιτήρησης ε, που έχει επιβάλει η Κροατία. Ε, υπάρχουν επίσης διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, στις οποίες βασιζόμαστε και από τις οποίες λαμβάνουμε και στοιχεία. Επίσης, δεν είναι θέμα της ε, Κομισιόν το πώς ε, φέρονται κάποιοι ε, αστυνομικοί. Θα πρέπει οι, κροατικές αρχές να λύσουν αυτό το θέμα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε τώρα στο σημείο 25, δηλαδή στα διάφορα. Δεν ε, βλέπω να υπάρχει κάτι στα διάφορα, άρα σημείο 26, 11 ε, Νοεμβρίου 2019 στις 3 ε, το απόγευμα μέχρι τις 6.30 στις Βρυξέλλες θα λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση, καθώς επίσης και την 12η Νοεμβρίου 2019, τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 και από τις 2.30 έως τις 6.30 πάλι στις Βρυξέλλες. Καλό σας βράδυ.